Έχοντας εγκρίνει την ημερήσια διάταξη, ας περάσουμε στο επόμενο σημείο. Την έγκριση δηλαδή των πρακτικών στις 26 Οκτωβρίου, 31 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Σημείο 4. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Those in the room remain silent. Όσοι παραμείνετε στην αίθουσα, να ησυχάσετε παρακαλώ. Προχωράμε στο σημείο υπαριθμών 4. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνη σε σχέση με το ρόλο του ΣΥΤΣΕΝ, Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είχα αποστείλει μία επιστολή στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Άστον, για μία ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΙΕΔ θα το συζητήσουμε από κοινού με τους συναδέλφους από τις Επιτροπές ΑΦΕΤ και ΣΕΝΤΕ. Καλωσορίσω τον κύριο Κριστόφ ε, Λιζέκ, αντιπρόεδρο της ΣΕΝΤΕ και από την ε, ΑΦΕΤ τον πρέσβη Πιέρ που είναι εκτελεστικός ε, σύμβουλος της ΕΙΕΔ και τον κύριο Σαλμή που είναι υπεύθυνος του ΣΥΤΣΕΝ, του Κοινού Κέντρου, ε, διευθυντής του ΣΥΤΣΕΝ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρήσεων. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον πρέσβη και μετά στον κύριο Σαλμή. Και μετά θα γίνει συζήτηση μετά από τις δύο εισηγήσεις. κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. επειδή νομίζω ότι ο πραγματικός σημερινός ήρωας είναι στο πλευρό μου. Είναι ο διευθυντή ε, του ΣΥΤΣΕΝ, του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι νομίζω ότι αυτά που θα σα πείτε θα σα ενδιαφέρουν. Παρακαλώ. Ησυχία παρακαλώ. Αυτό θα μας βοηθήσει. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μιλάω πιο δυνατά και πιο κοντά στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα θα σας τα πει ο συνάδελφός μου, η ε, Κασάλμη, η Διευθύντρια, και θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι σχέσεις που είχαμε μεταξύ της εξωτερικής διάστασης και της εσωτερικής διάστασης της πολιτικής ασφάλειας που έχουμε. Και αυτό ήταν το ευρύτερο ερώτημα που θέσατε. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στην Ιλκα, η οποία θα επισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ΣΥΤΣΕΝ. Γνωρίζουμε όλοι και είναι περιττό να επαναλάβω ότι στον τομέα της ασφάλειας βασικό είναι φυσικά να υπάρχει συνοχή, συντονισμός μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης των ε, ευρωπαϊκών δράσεων όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να κτίσουμε ένα τείχο μεταξύ των δύο, διότι είναι αλληλένδετες στον κόσμο που αντιμετωπίζουμε σήμερα και το γνωρίζουμε είτε όταν πρόκειται να αυξήσουμε τις προσπαθειές μας για να αντιμετωπίσουμε την αντιτρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα ή για να αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση και το λαθρεμπόριο που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναφέρω λίγες από τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας. Άλλωστε πρέπει να δούμε και την εξωτερική διάσταση αυτών των απειλών. Αυτό είναι προφανές. Βλέπουμε καθημερινά αυτές τις απειλές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να συνεργαζόμαστε στενά με τα διάφορα κράτη-μέλη με βάση τις διμερείς μας σχέσεις και πρέπει να συνδυάζουμε τους στόχους αυτών των δράσεων των κρατών μελών με τους στόχους του πολιτικού μας διαλόγου με τις τρίτες χώρες. Την εξωτερική βοήθεια που παρέχουμε σε αυτές τις χώρες και επίσης τις αποστολές για διαχείριση των κρίσεων. Όποια και αν είναι τα σχέδια δράση που πρέπει να αναλάβουμε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν ε, συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ο σωστό δρόμος. Όχι μόνο με τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαζόμαστε πολύ στενά, αλλά και με την Επιτροπή. Και με την Επιτροπή λοιπόν ήδη έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τον συντονισμό των προσπαθειών μας, όπως και τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων. Όπως γνωρίζετε, μόλις υιοθετήσαμε δύο στρατηγικές ε, προτεραιότητες για το κέρας της Αφρικής και το Σαχέλ και, το Σαχέλ και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις ενέργειες, της δράσης και να υλοποιήσουμε τα προγράμματα μέσω εκείνου το οποίο ονομάζουμε ενοποιημένη ή ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, λοιπόν, η εξωτερική και η εσωτερική διάσταση αποτελούν μέρος της καθημερινής μας δραστηριότητας. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα των ε, αρχικών σταδίων που καλύψουν. Ε, Οι εκπρόσωποι της ISS ε, έχουν την έδρα τους, αν θέλετε, και συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, που έχουν να κάνουν με θέματα εσωτερικής ασφάλειας όπως Κοζίκα, ΕΞ και ούτω καθεξής. Και η ΕΣ επίση, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, εκπροσωπείται σε επίπεδο διευθυντών στην Υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας που πρόσφατα δημιουργήθηκε υπό την διεύθυνση της Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Και με, με τα χαρά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η υπηρεσία μας πρόκειται να δημιουργήσει και άλλη ομάδα μεταξύ υπηρεσιών όσον αφορά ε, την εξωτερική διάσταση, την εξωτερική ασφάλεια. Και η υπηρεσία μας θα προεδρεύσει αυτές τις υπηρεσίες και θα εργάζεται πολύ στενά με την Επιτροπή. Ένα κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πρόκειται να ε, δημοσιοποιηθεί στην αρχή του επομένου μήνα που θα διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ του CSDP ε, και του τομέα της ελευθερίας, ε, ασφάλειας και δικαιοσύνης αναζητώντας συνεργασία μεταξύ των σημαντικών παραγόντων για να δουν ποια διασύνδεση μεταξύ των πολιτικών μπορεί να υπάρξει ώστε να καταλήξουμε σε συντονισμένες ενέργειες στο μέτρο του δυνατού. Αφού λοιπόν δημοσιευθεί και υποβληθεί αυτό το έγγραφο στο PSC, θα υπάρξει μια κοινή συνάντηση του PSC και του COSI. Νομίζω ότι είναι η πρώτη συνάντηση αυτής της μορφής που σχεδιάστηκε για αρχές Ιουνίου και θα συζητήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί η διάσταση στον τομέα της ασφάλειας, η εσωτερική διάσταση και η εξωτερική διάσταση ήδη και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε ήδη στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος στο Χόλμης έχει γίνει σημαντική δουλειά με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των πολιτικών αποστολών και ε, της ε, ελευθερίας, ασφάλειας και της δικαιοσύνης κυρίως όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπόλ και όσον αφορά τις διάφορες πολιτικές αποστολές τις οποίες έχουμε οργανώσει ε, στον τομέα ε, της πολιτικής προστασίας, ε, χωροφυλακή, αστυνομία σε διάφορες περιοχές όπως το Κόσοβο ή το Αφγανιστάν. Επίσης, σκοπεύουμε σε αυτή την κοινή συνάντηση να αναζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης αυτή Τη της ε, συνοχής εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής όταν έχουμε θέματα αντιτρομοκρατίας και όταν έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που έχει γίνει μία από τις βασικές προτεραιότητες ε, της ε, ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της ασφάλειας. Οφείλουμε και θα αναλάβουμε πολλές πρωτοβουλίες σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα αλλά θα προχωρήσουμε περαιτέρω και βεβαίω όλες οι προτεραιότητε στον τομέα της ασφάλειας όπως ορίζονται και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας ή στην ε, Στρατηγική εσωτερική Ασφάλειας θα επεκταθούν ε, σε αυτές τις κοινέ δράσεις που αναλαμβάνουμε όλοι εμείς ε, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Επίσης, διερευνούμε τη δυνατότητα ενίσχυσης ορισμένων ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών μας που έχουν προτεραιότητες για θέματα ασφάλειας σε μια προσπάθεια ενίσχυσης αυτών με εμπειρογνώμονες όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας και θα γίνουμε κάπως ε, σύνδεσμοι ε, σε θέματα που έχουν σχέση με την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Δεν θα ήθελα όμως να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση χωρίς να επαναλάβω ε, την δέσμευσή μας σε αυτό το τομέα και να απογραμμίσω την ανάγκη παγίωσης του κράτους δικαίου, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου που αποτελούν τις βασικές αξίες όλων των ευρωπαϊκών προσπαθειών για τη διατήρηση της ειρήνης, ε, για την αποτροπή των συγκρούσεων και για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας δεν είναι μόνο υποχρέωση βάση των συνδικών, αλλά είναι και προσωπική μου πεποίθηση ότι είναι πολύ σημαντική και επίσης είναι πεποίθηση της ύπαρξης εκπροσώπου. Θα ήθελα να σα πω ότι οι περισσότερε αποστολέ μα είναι πολιτικές, ε, είτε όσον αφορά το κράτος δικαίου, είτε τον τομέα της μεταρρύθμισης του τομέα τη ασφάλεια. Συνήθω εστιάζονται στην ανάγκη και στην υποστήριξη ε, των χωρών για την επαναλειτουργία του τομέα της ασφάλειάς τους σύμφωνα με δημοκρατικούς κανόνες και τις αρχές της υγιούς διακυβέρνησης. Αυτή είναι δέσμευσή μας και τους επόμενους μήνες θα πρέπει να οργανώσουμε νέες αποστολές ε, όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ασφάλεια και την ε, αναμόρφωση αυτόν τον τομέα. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εκεί και θα δώσω για να πάει, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βιλμό. Όπως προβλέπετε τώρα, έχουμε τον κύριο Σάλμη. Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι ως συνήθως έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη και για σήμερα το απόγευμα αρκετά σημεία στην ημερήσια διάταξη και γι' αυτό ζητώ τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να συντομευσουμε εξι 6-7 λεπτά για την παρουσίαση θα ε, ήθελα να χρησιμοποιήσετε για να έχουμε χρόνο και για τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ο κύριος Σάλμη θα μπορούσα να σας βοηθήσω και να μην πω κουβέντα καθώς προέρχομαι από το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων και να κρατήσω το στόμα μου σφραγισμένο. Όμως θα ήθελα να κάνω αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Υπάρχουν διάφορες φήμες ε, και παρανοήσεις στις Βρυξέλλες για το ρόλο του κοινού κέντρου επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα ε, κάπως ε, να διαλευκάνω αυτό το θέμα. Καταρχήν να μιλήσω για την αποστολή μας, για τα καθήκοντά μας και για τη λειτουργία μας καθώς και ορισμένα από τα αποτελέσματα του κοινού κέντρου επιχειρήσεων. Ξεκινώ με την αποστολή μας για να μπορέσουμε να έχουμε μια ασφαλή Ευρώπη σε ένα ε, παγκόσμιο πλαίσιο, όπως αναφέρεται στη στρατηγική μας, χρειαζόμαστε τις σωστές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να ε, λαμβάνουμε τις σωστέ αποφάσεις πολιτικής και για θέματα εσωτερική και για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η αποστολή του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το να παρέχει ανάλυση των πληροφοριών ε, εγκαίρως προς την ύπατη εκπρόσωπο την κυρία Άστον και προς όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο πλαίσιο της ε, ΚΕΠΑ και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας το κοινό κέντρο επιχειρήσεων να διεξάγει την αποστολή της παρακολουθώντας διεθνή γεγονότα ε, επί 24 ώρου βάσεως και καθημερινά χωρίς να διακόπτουμε καθόλου. Μας απασχολούν τομείς όπως η τρομοκρατία, η διάδοση ε, των μέσων μαζικής, των όπλων μαζικής καταστροφής ε, και άλλα συναφή θέματα. Θα σας πω δύο λόγια για το ιστορικό της δραστηριότητα του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων. Η δημιουργία του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων έχει άμεση σχέση με την ε, κοινή πολιτική ε, ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες διαχείρισης κρίσεων και η δυνατότητα αποστολών ε, στρατιωτικών πολιτικού και μη στρατιωτικού χαρακτήρα, κατέστησαν σαφέ ότι χρειάζεται ανάληψη δράση σε αυτό το τομέα. Από τα γεγονότα της 11 ε, Σεπτεμβρίου του 2001, καταλάβαμε ότι χρειάζεται μια ανάλυση των πληροφοριών εγκαίρως για να υποστηρίξουμε τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το 2002 δημιουργήθηκε το Κοινό Κέντρο Επιχείρησεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω Γενική Γραμματεία που υπόκειτο στον είπα το εκπρόσωπο το 2005 ενισχύθηκε το κοινό κέντρο επιχειρήσεων με μια ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπάστησαν από την ομάδα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να παρέχονται οι επιχειρήσεις που παρέχονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, δηλαδή ε, υπηρεσίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με βάση πληροφορίες από τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Από το 2007 το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων συνεργάζεται με την Διεύθυνση Πληροφοριών ε, του, της μονάδας ε, μη στρατιωτικής ε, δράσης και τα προϊόντα τα οποία εμείς παράγουμε παράγονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών. Τέλος, με τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας τον Σεπτέμβριο του 2009, το κέντρο επιχειρήσεων πέρασε στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ ε, της, της της κυρίας Άστον ε, και πέρασε το 2011 στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Στις 26 Ιουλίου του 2010 πέρασε στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, καθήκοντά μας ε, είναι η ανάλυση κινδύνου και η, εξέλιξη, η παρακολούθηση και ανάλυση ε, πληροφοριών. Συνεχίζουμε τα καθήκοντα αυτά και αναλύουμε τις πληροφορίες. Παράγουμε εγκαίρως εκθέσεις για τη διαχείριση κρίσεων και Προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τις ώρες λειτουργίας και εκτός δηλαδή των ωρών εργασίας. Σε επίγουσες καταστάσεις έχουμε επί 24 ώρου βάσεως παρακολούθηση. Έχουμε μονάδες ανάλυσης, μονάδες ε, επικοινωνιών. Έχουμε επίση ε, και συμφωνίες με το ε, σύστημα πλοήγησης μέσω δορυφόρου για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους. Τα συστήματα πληροφοριών, όπως καταλαβαίνουν και οι απλοί άνθρωποι, έχουν σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται για απόρριτα θέματα. Αυτό ε, δεν αληθεύει όμως ε, επακριβώς, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από δικές μας ε, αποστολές και πληροφορίες και από τις πληροφορίες που μας δίνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών. Και τονίζω ότι το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μια υπηρεσία ασφαλείας η υπηρεσία πληροφοριών όπως αυτές που λειτουργούν στα κράτη-μέλη και κατά τη γνώμη μου θα απαιτεί το αλλαγή στη συνθήκη και τεράστια πολιτιστική αλλαγή αν υπήρχε μια κατάσταση στην οποία θα προσπαθούσε το κοινό κέντρο επιχειρήσεων να γίνει τέτοιου είδους φορές, δηλαδή ανάλογος με τα κέντρα πληροφοριών των κρατών μελών αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ρόλος των κρατών μελών ε, και είναι θέματα εθνικής ασφάλειας οι πληροφορίες. Εμείς, όπως σας είπα, παρέχουμε ανάλυση πληροφοριών σε στρατηγικό επίπεδο για να βοηθήσουμε τη λήψη αποφάσεων και δεν παρέχουμε πληροφορίες ε, επιχειρησιακού χαρακτήρα όπως ε, τα οι υπηρεσίε πληροφοριών των κρατών μελών. Αυτέ ήταν οι αρχικέ μου παρατηρήσει, κύριε Πρόεδρε. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σάλμη. Τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Λίζεκ, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ. Έχετε το λόγο κύριε Λίζεκ. Θα μιλήσω πολωνικά. Έτσι θα μιλήσω γρηγορότερα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για αυτή τη συνάντηση, διότι σήμερα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας είναι θέματα που μας απασχολούν όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που οργάνωσε αυτή τη συζήτηση γιατί τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικά μέσα στα πλαίσια του, της κυβερνοτρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και ούτω καθεξής. Θα ήθελα όμως να σας ε, προκαλέσω κάπως κύριε Δευθυντά και κύριε Πρέσβη διότι μας μιλήσατε για την άποψή σας για ευρωπαϊκά θέματα πληροφοριών. Αυτό συζητήθηκε και από την Επιτροπή. Θα ήθελα όμως τη δική σας γνώμη. Όχι μόνο επειδή είπατε ότι ο δικός σας φορέας δεν είναι ένας κλασικός φορέας ε, πληροφοριών, αλλά πιστεύετε ότι σήμερα χρειάζεται ένας τέτοιος φορέας. Έχει λόγο ύπαρξης, έχει νόημα να προσδώσετε αυτό το χαρακτήρα στο φορέα σας, δηλαδή να είναι ένας, μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών. Οπωσδήποτε χρειάζεται συνεργασία, συνεργασία με άλλους φορείς όπως τη Europol, τη Frontex, ιδιαίτερα σχετικά με τις αποστολές και πά. Και επιπρόσθετα θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ της δικής σας, του δικού σας φορέα και άλλων υπηρεσιών πληροφοριών ανά τον κόσμο. Δεν μιλώ μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Σας ευχαριστώ τα μέλη ζήτησαν το λόγο, δύο λεπτά ο καθένας έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος. Η κυρία Ιντβελτ καταρχήν. Ευχαριστώ. Καταρχήν χαίρομαι ιδιαίτερα διότι διοργανώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Είναι κάτι που το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό, το έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Θα επικεντρωθώ στο θέμα του δημοκρατικού ελέγχου και εποπτείας γιατί εδώ και πολλά χρόνια ακούσαμε, ακούγαμε για το Σίτζεν, δεν ε, είχε παραδεχτεί κανένα στην ύπαρξή του και τώρα φαίνεται σαν ένα μόρφωμα που αναδύεται από την ομίχλη. Εσείς είπατε ότι δεν είναι μια επιχειρησιακή οργάνωση, ότι βρίσκεστε υπό την Βαρόνη Άστον αλλά εάν είναι, έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Ίσως αυτό είναι θετικό γιατί νομίζω ότι η συνεργασία σε αυτό το τομέα είναι απόλυτα αναγκαία αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να οργανώνουμε και τη δημοκρατική εποπτεία. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συσταθεί μια τέτοια υποδομή, δηλαδή μια επιτροπή μέσα στα πλαίσια ε, θεμάτων ασφαλείας και διεκπαιρέωσης θεμάτων ασφαλείας. Θεωρώ ότι έχουμε θέματα επιτάπητος που θα συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών για λόγους που είναι μυστηριώδεις ε, σε μένα, γιατί αν θέλουμε πραγματικά να εποπτεύσουμε, ε, να προβάλλουμε ε, τον, ε, τη δημοκρατική εποπτεία, αυτό το θέμα θα έπρεπε να ήταν και κλεισμένο των θύρων. Κλείνει τώρα ο κατάλογος έτσι ώστε να έχετε χρόνο όλοι. Ο κύριος Άλβαρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων. Χαίρομαι λοιπόν που είσαστε εδώ. Όπω είπε και η κυρία Ινβέλτ, θέλαμε μια τέτοια συνάντηση εδώ και καιρό. Μίλησε και ο κύριος Δημό για το θέμα μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το ακούμε και από, από το ΕΛΚ και από τους σοσιαλιστές σχετικά με το τι θα μπορούσε να είναι και ε, τι είδους απέτηση θα μπορούσαμε να έχουμε για τη δημιουργία ενός τέτοιου ευρωπαϊκού ε, ε, φορέα. Δεν έχω κάποια τελική θέση εγώ από την πλευρά του Άριντε. Ξέρω ότι και πολλά κράτη-μέλη έχουν πολλές επιφυλάξεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου επιχειρησιακού κέντρου και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο σε σχέση με το Συμβούλιο. Ο κ. Δεκέρκοφ ε, είπε προσφάτως ότι υπό την ε, η ηγεσία του θα μπορούσε ε, να συνδυαστούν, θα μπορούσαν να συνδυαστούν ε, δράσεις καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Εμάς μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο οι διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουζουτήλ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερις πολύ σαφείς ερωτήσεις προς τον κύριο Σάλμη. Το CITCEN, το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων, συνεργάζεται με φορείς όπως η Frontex, που έχει επίσης το δικό της κέντρο επιχειρήσεων, ή με την Europol. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν ε, τα στοιχεία πληροφοριών τα οποία παίρνετε εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων. Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων ε, έχει, μοιράζεται πληροφορίες ε, με τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τέταρτον βλέπετε το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων να έχει κάποιο ρόλο ε, σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ένα πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδότησης τρομοκρατίας TFTP σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ευρωπαϊκό σύστημα ENPI. Η κυρία Ρομέρο Λόπες, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι, ποιες είναι οι τρομοκρατικές απειλές που γνωρίζει τώρα η Ευρώπη σύμφωνα με την πείρα σας που αποτελούν ε, αναπόσπαστο τμήμα εργασιών αυτού του κέντρου. Και δεύτερον, επειδή είπατε ότι οι έρευνες είναι ίδιες έρευνες, που συλλέγουν τις ε, πληροφορίες των στρατιωτικών υπηρεσιών είναι γεγονός ότι εάν ε, οι υπηρεσίες πληροφοριών κάθε χώρας δεν ε, συντονίζονται είναι δυσπρόσιτες, τότε υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη συντονισμού στα κράτη-μέλη. Αυτό το είδαμε με, τις 16, με τους 16 φορείς στις ΗΠΑ που δεν μπόρεσαν να κατατροπώσουν την τρομοκρατία. Το ίδιο ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω κατά πόσο στα κράτη-μέλη υπάρχει αυτή η έλλειψη συντονισμού. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, Πώς το βλέπετε σε επίπεδο ανάλυσης, δηλαδή μπορεί αυτό το κέντρο να έχει πληροφορίες, συντονισμένες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, όχι σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο ανάλυσης. θα μπορούσε να υπάρξει να προωθηθεί αυτό το εγχείρημα συντονισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε τελικά την ευκαιρία να μπορέσουμε διεξοδικά να συζητήσουμε αυτά τα θέματα ε, σχετικά με το ρόλο του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιολογεί τις πληροφορίες ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρήσεων. Θα με ενδιαφέρε να μάθω ποια είναι η σχέση σας με τη Europol και τη Eurojust. Πώς ανταλλάσσετε πληροφορίες με αυτούς τους οργανισμούς. Πώς γίνεται η επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τα στοιχεία της Europol. Και ε, ιδιαίτερα με ενδιαφέρει το θέμα του ε, ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου στο στον οποίο υπόκειστε. Σε ποιο κοινοβούλιο και σε ποιο κοινοβουλευτικό έλεγχο υπόκειστε. Στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολύ αυστηρές διατάξεις για τον έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών σε πολλές περιπτώσεις σήμερα υπό την έννοια καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, δίδεται η δυνατότητα να συμβεί οτιδήποτε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει με την απλή δικαστική αστυνομική συνεργασία όπως αυτό που κάνει η Europol και η Eurojust. Γι' αυτό θέτω εγώ το ερώτημα, το πώς βλέπετε το κοινό πλαίσιο της συνεργασίας σας με τη Europol και τη Eurojust και ποιος είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος τον οποίο υπόκειστε. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω για τα θέματα καταπολέμησης της ε, εγκληματικότητας ε, και τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο εξωτερικό φορέα γιατί πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψη σε αυτόν. Κύριε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο πρόεδρος κ. υπογράμμιζε τη σημασία του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών κανόνων. Μπορεί να μας πει αν γνωρίζει τι συνέβη ε, στις ε, διατλαντικές νομικές συζητήσεις ε, που ξεκίνησαν από την πλευρά της Αμερικής, αν δεν απατώμε, υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Και ας το πω κάπως απλά, είχαν ως αντικείμενο να κάνουν την Ευρώπη να αποδεχθεί ότι η απλή ε, ε, ποινική δικαιοδοσία δεν ίσχυε για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας όπως οι απαγωγές κτλ. Μπορεί να μας πει, διότι δεν έχω ακούσει τι έχει συμβεί με αυτά τα θέματα, τι συμβαίνει δηλαδή κυρίως υπό το φως της ε, του γεγονότος ότι ο πρόεδρος Ομπάμα συνεχίζει να έχει τις επιτροπές, στρατηγικές επιτροπές ε, ε, στο Γκαντάναμο. Then, Mrs. Lunacek, two minutes. Thank you. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω συνέχεια στα όσα είπαν οι συνάδελφοι για το θέμα της Δημοκρατού Ελέγχου. Και ω μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εξεπλάγει που βλέπω ότι εδώ γίνεται αυτή η συζήτηση ε, του κέντρου επιχειρήσεων, αλλά αυτό αποτελεί μέρο ε, τη εξωτερική υπηρεσία. εξωτερικής υπηρεσίας. Και είναι ενδιαφέρον που γίνεται εδώ η συζήτηση και όχι στα πλαίσια τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν και στι δύο επιτροπέ. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά όσον αφορά ε, το ερώτημα που έκαναν άλλοι, αυτή η ιδέα του κ. Κέρκοβ ίσως να έχουμε ένα ε, κεντρικό οργανισμό μεταξύ ε, Ουβροπόλ και ε, του Κέντρου Επιχειρήσεων. Πόσο προσωπικό έχει αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα οριζόντια και γραφικά θέματα τα οποία σας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Και ποια είναι η διαφορά με τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Έχετε δικές σας πηγές. Αναφέρατε ορισμένε ορισμένες πηγές που σας δίνουν πληροφορίες. Αλλά προσπαθείτε να έχετε και δικές σας πηγές πληροφόρησης. Δημιουργείτε δικές σας, δικές σας πηγές πληροφόρησης. Και για να το ποσοτικοποιήσουμε αν θέλετε. Πόσο ποσοστό της καθημερινής δουλειάς της ΣΥΤΣΕΝ είναι δουλειά η οποία αφορά την αντιτρομοκρατία και πώς, πώς, το ποσοστό των δραστηριοτήτων σας για την αντιτρομοκρατία και ποιο ποσοστό αφορά τα άλλα θέματα. Τι σημασία δίνεται όσον αφορά ε, την αντιτρομοκρατία, πώς, πώς το συνδέεται με την ε, ε, πολιτική ασφάλειας. Κύριε Μπρόγκ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχήν για το κέντρο επιχειρήσεων, το CITSEN μπορείτε να αφαιρθείτε σε ένα συμβάν ή σε πολλά συμβάντα που μπορέσατε εσείς να προβλέψετε από τις ανοιχτές πηγές που έχετε και πότε ε, αντιληφθήκατε ε, τις αναταραχές στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή πολύ πριν από ε, εμάς. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεύτερον, υπήρξαν ορισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις που μπορέσατε να αποτρέψετε. Ίσως δεν θέλετε να μας ονομάσετε ποιες, αλλά θα μπορούσατε να μας πείτε κατά πόσον αυτό συνέβη, μπορέσατε να σας αποτρέψετε. Ένα άλλο θέμα όσον αφορά το αιώνιο θέμα της ελευθερίας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης. Πάντοτε σκέφτομαι το εξής. Η ελευθερία σημαίνει πολλά περισσότερα όσον αφορά ε, την, ε, την, την καταπάτηση των ποινικών συστημάτων των κρατών μελών και κατά πόσον υπάρχει κάποια έννοια που έχετε δώσει στο θέμα του εγκλήματος. Το θέμα είναι ότι ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης μπορούν να φυλακιστούν άτομα σε άλλες χώρες αναμένοντας να δικαστούν. Σταματάω εδώ γιατί περάσαν τα δύο λεπτά μου. Ευχαριστώ. Ο, κύριο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ καταρχήν θα ήθελα ορισμένα αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που προείπε και η κυρία Λούνατζεκ. Δηλαδή πόσο προσωπικό διαθέτεται, πόσοι είναι εμπειρογνώμονες, πόσοι προέρχονται από ε, τα εθνικά κράτη-μέλη, πόσοι είναι καθαρά δικοί σας υπάλληλοι. Σε σχέση με τον επιχειρησιακό χαρακτήρα του φορέα, επειδή δεν είμαι εμπειρογνώμων, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η οριοθέτηση μεταξύ ε, αναλυτικού χαρακτήρα και επιχειρησιακού χαρακτήρα. Γιατί εσείς μιλήσατε για επιχειρησιακό επιχειρησιακό χαρακτήρα πέρα από τα θέματα επικοινωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς προσλαμβάνει ο φορέας αυτό τον επιχειρησιακό χαρακτήρα. Γιατί εάν ε, εργάζεστε με ε, δευτερογενείς πηγές, το ζήτημα είναι διαφορετικό. Ως προς τις αποστολές, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο ε, έχετε ένα σύστημα σαν το κέντρο παροχής πληροφοριών μέσω δορυφόρου. Με βάση τα πρόσφατα γεγονότα της Λιβύης και τις εκθέσεις σας, γιατί ίσως γνωρίζετε ότι εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή έγγραφα εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα της Λιβύης και ζήτησα από εσά να ε, εξετάσω ορισμένα έγγραφα τα οποία δεν μου χορηγήθηκαν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι πηγές άμεσες ή έμεσες χρησιμοποιήσατε και κατά πόσο υπάρχουν ειδικέ αναλύσεις με βάση συγκεκριμένες πηγές ή βασίζεστε στις Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Η κυρία Χάνκης. Two minutes, please. Για δύο λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Σάλμη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με ενδιαφέρει η σχέση του ΣΥΤΚΕΝ, με τα κρατη διότι ξέρουμε ότι υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας της συνθήκης της Λισαβόνας, ότι δηλαδή τα θέματα ασφαλείας είναι καθαρά εθνικής ευθύνης. Αυτό είναι πρόβλημα για το ΣΥΤΤΣΕΝ. Θα υπήρχε πρόβλημα πραγματικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Και θα, πώς θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα δραστήριο στα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ίσως αυτός ο συσχετισμός λοιπόν. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πολύ σύντομη. Πολύ συχνά μιλάμε για το θέμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον θα πρέπει να έχει τη δική της υπηρεσία πληροφοριών. Θα ήθελα την δική σας άποψη. Δηλαδή είναι μια ερώτηση μελλοντολογίας καθαρά. Ευχαριστούμε κύριε Χάκης. Αρκετά σημεία εθίγησαν από μέλη της ΑΦΕΤ και της ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ γιατί τηρήσατε το χρόνο και υποβάλατε συγκεκριμένες ερωτήσεις, γι' αυτό θα πρότεινα να έχουμε ένα διπλό γύρο ε, απαντήσεων. Κύριε Βημό ή ο κύριος Σάλμι αν προτιμά να αρχίσει σε σχέση με όσα θέματα εφήγησαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που έγιναν. Πρώτα απ' όλα πώς προχωράμε και πώς βλέπω το μέλλον ε, του τομέα των πληροφοριών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες και με ορισμένους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τρίτον, οι δημοκρατικές βάσεις ε, του ΣΥΤΣΕΝ, του κέντρου. Και κατόπιν θα απαντήσω σε πιο συγκεκριμένα ερωτήματα όσον αφορά το προσωπικό και τα λοιπά, σχετικά με το κέντρο επιχειρήσεων και πώς ε, κάνουμε τις δραστηριότητες μας. Λοιπόν, ξεκινάω με το εξής. Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον ε, όσον αφορά τη συνεργασία στο δομέα της πληροφόρηση, των πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ε, ε, εναρτήριε παρατηρήσει μου είχα πει ότι πιστεύω ότι τα θέματα τη εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης ε, των πληροφοριών είναι δικαιοδοσία των κρατών μελών. Και ρωτήθηκε τι αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν εάν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό οργανισμός πληροφοριών Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί στις συνθήκες, δηλαδή να γίνει τροποποίηση των συνθήκων. Έτσι πιστεύω, διότι, το υπογραμμίζω, η εθνική ασφάλεια είναι στις αρμοδιότητε των κρατών μελών. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον, ούτε μεσοπρόθεσμα θα έλεγα, είναι δυνατό να υπάρξει, ίσως και όχι μακροπρόθεσμα. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή λοιπόν Υπηρεσία Πληροφοριών. Προσωπικά προτιμώ μια στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών που υπάρχουν σε πολλά μέτωπα. Και αυτό είναι ο τρόπος που βλέπω για το μέλλον. Τώρα είναι και θέμα πόρων. Ήδη τα κράτη-μέλη έχουν τέτοιε δραστηριότητε και πρέπει να σκεφτούμε τι προστιθέμενη αξία θα παρουσίαζε ε, μία υπηρεσία επιχειρήσεων. Επίσης, μου είπαν ότι υπάρχει μια μονάδα επιχειρήσεων στην ΣΥΤΣΕΝ. Ναι, υπάρχει. Αλλά ασχολείται μόνο με θέματα απόκρισης στην κρίση. Ε, είναι ένα σύστημα το οποίο έχουμε που δεν αφορά όμως ε, τις πληροφορίες. Αφορά μόνο τις κρίσεις και συμμετέχει ε, στις πληροφορίες, ανοιχτές πληροφορίες, αναλύει ε, τις ε, πηγές, αλλά οι δικές μας πηγές διαδιευθύνονται από ΣΥΤΣΕΝ. Βασίζουμε τις εκτιμήσεις μας την εργασία μας στις ανοιχτές πηγές, στην παρακολούθηση των μέσων, των αποστολών, στις πληροφορίες των αντιπροσωπιών και στην ροή των πληροφοριών που μας δίνουν οι υπηρεσίες των κρατών μελών. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε πληροφορίες εμείς το ΣΥΤΣΕΝ δεν είναι ένα κέντρο το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες μόνο του. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές. Τώρα, οι σχέσεις με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους ή με τις τρίτες χώρες συνεργαζόμαστε όταν υπάρχουν συμφωνίες ασφάλειας με την Ελβετία, την Ορβηγία στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Αυτοί είναι οι κύριοι εταίρες μας. Κατά η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται μεταξύ κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, πολλοί ρώτησαν ποια είναι η σχέση μεταξύ Frontex, Europol και CITSEN μεταξύ άλλων. Θα έλεγα, για παράδειγμα, αν η Frontex, ή μάλλον, ναι, συνεργαζόμαστε με τη Frontex, έχουμε ορισμένε ρυθμίσει και συμφωνίε για ανταλλαγή πληροφοριών, όπω και με την Europol. Ένα από τα προϊόντα στα οποία, τα οποία δημιουργούμε μαζί με την Europol είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε T-SAT, ένα έγγραφο που από κοινού βγαίνει. Επίσης, το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως ε, το ζήτημα των δεδομένων. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι εμείς δεν συλλέγουμε δεδομένα ή πληροφορίες για τα άτομα. Εμείς κάνουμε στρατηγικές αναλύσεις. Δεν έχουμε λοιπόν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα καθόλου και κατά τη γνώμη μου αυτό δεν χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας. Τώρα, η δημοκρατική παρακολούθηση του ΣΥΤΣΕΝ είναι κάτι που αναπόκειται σε εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Να αποφασίσουν κατά πόσον το θέλουν. Ανάλογα με τα κράτη-μέλη, τα συστήματα είναι διαφορετικά. Και αν δεν απατώμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μία έρευνα των διαφόρων συστημάτων, ζητώντας τα κράτη-μέλη να δώσουν πληροφορίες για το πώς γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχει σαφή διαφορά ανάμεσα στις υπηρεσίες των κρατών μελών και τη ΣΥΤΣΕΝ επειδή εμείς δεν συλλέγουμε από μόνοι μας πληροφορίες. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, όσον αφορά το δικό μας το σύστημα και τα συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και από ό,τι γνωρίζω ε, τα κράτη-μέλη έχουν εντελώς διαφορετικά συστήματα. Με άλλ, το κάθε, η κάθε χώρα έχει το δικό της τον τρόπο για να παρακολουθεί ε, την ασφάλεια της χώρας. Επίσης έγιναν ερωτήσεις σχετικά με το ε, προσωπικό. Έχουμε 100 και λίγο περισσότερους προς το παρόν. Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι είναι οι εμπειρογνώμονες και ποιοι είναι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω μαζί μου τα ακριβή στοιχεία, αλλά η αναλογία είναι 70-30 περίπου. Αλλά αυτό το λέω, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία. Τώρα, το ποσοστό των δραστηριοτήτων μας ε, που συμβάλλουν ε, στο ΣΥΤΙ, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας το πω. Αυτό εξαρτάται ο οργανισμό μας είναι σχετικά μικρός. Σε περίπτωση όπω η Λιβύη, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη περιοχή της Μέση ανατολή εκεί αφιερώνουμε περισσότερους πόρου μας και το προσωπικό μα ασχολείται κυρίως με αυτά τα θέματα. Πάλι όμως, αν χρειαστούν περισσότερε δραστηριότητε, θα κατανείμουμε διαφορετικά τους πόρου μα. Δεν μπορώ να σα απαντήσω λοιπόν αναφέροντας ποσοστά. Επίσης μου ζήτησαν ποια είναι τα ουσιαστικά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Σίγουρα η αντιτρομοκρατία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας, αλλά ανάλογα και με τα ε, hot spots που υπάρχουν, φυσικά εστιαζόμαστε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση και στη Βόρεια Αφρική και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν είναι το θέμα της μη διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής που αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης. Επίσης μου ζήτησαν ποιες είναι οι τρομοκρατικές απειλές για την Ευρώπη. Αυτό εξαρτάται από ε, ε, κράτος σε κράτος. <clears throat> Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι συλλογικά να εξετάζουμε την κατάσταση των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης και να εκτιμήσουμε, για παράδειγμα, ε, τα προβλήματα που μπορεί να έχουν στα ταξίδια ορισμένα άτομα, σε ορισμένα κράτη-μέλη και προειδοποιούμε για τους τυχόν κινδύνους. Πρόεδρο, εάν ο κύριος Πρέσβης θέλει να συνεχίσει, ε, θα δω μήπως, ε, μήπως μπορεί να καλύψει μένα ερωτήματα τα οποία δεν κάλυψα εγώ. Βεβαίως, ε, κύριε Μπεμό, ευχαριστώ. Θα προσθέσω λίγες παρατηρήσεις στα όσα είπε ίδιο ο συνάδελφος. η γενική ιδέα την οποία διατυπώσατε πολύ από εσά, δηλαδή κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας ή Προφοριών. Ήδη απαντήθηκε αυτή η ερώτηση, αλλά θα μπορούσα ίσως να προσθέσω μερικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι εξή. Αυτό δεν αφορά μόνο τα χρήματα, αλλά πώς θα εκπαιδεύσουμε τα σωστά άτομα. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο πληροφοριών, αυτό χρειάζεται χρόνο, πολύ χρόνο και επίσης πρέπει να βρείτε τους σωστούς ανθρώπους αν θέλετε να είσαστε αποδοτικοί. Τρίτον, είναι και θέμα της επικάλυψη. Όπω είπα, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν τις ικανότητες αυτές και τις υπηρεσίες αυτές και θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό το θέμα, διότι έγινε μια παρατήρηση σχετικά με το συντονισμό και τη συνεργασία στο εσωτερικό κάθε χώρας. Φαντάζεστε λοιπόν αν προσθέσουμε και άλλο επίπεδο ε, δικτύου πληροφοριών πέραν εκείνων που υπάρχουν ήδη. Νομίζω ότι αυτό είναι από τους λόγους που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και μέχρι τώρα, όπως υπόθηκε, οι συνθήκες δεν έχουν προβλέψει κάτι τέτοιο. Τώρα, αναφορικά με το συντονισμό στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα εντός των κρατών μελών. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ε, Βλέπετε τι έγινε στι Ηνωμένε Πολιτείε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έγιναν πολλές προσπάθειες ε, για να συντονιστούν οι εθνικοί οργανισμοί έγιναν μεταρρυθμίσεις εδώ και εκεί και σε κάθε κράτος μέλος έγιναν μεταρρυθμίσεις και καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες και από πλευρά των Αμερικανών φίλων δεν είμαι βέβαιος ότι οι προσπάθειες πάντοτε υπήρξαν αποτελεσματικές, αλλά όλοι κατάλαβαν το πρόβλημα ήταν μείζον και ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ΣΥΤΣΕΝ είναι ότι στο επίπεδο της Ευρώπης προσπαθήσαμε να συντονιστούμε κατά κάποιο τρόπο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό μπορεί να μας ωφελήσει όλους όταν πρέπει να συσχετίσετε την εσωτερική με την εξωτερική διάσταση. Τέθηκε το ερώτημα γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, διότι εδώ αυτό ενέχει ένα εξωτερικό στοιχείο. Το έγκλημα δεν σταματάει στα σύνορα, αλλά επεκτείνεται παντού, είναι διασυνοριακό το έγκλημα και μερικές φορές μπορεί να έχει σημαντικές διασυνδέσεις με την τρομοκρατία. Και όλα αυτά λοιπόν όλο και περισσότερο διασυνδέονται και μας δείχνουν ότι χρειάζεται όχι μόνο να περάσουμε από το μεγάλο έγκλημα στη δρομοκρατία, αλλά και από την εσωτερική ασφάλεια στην εξωτερική ασφάλεια. Υπάρχει διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο εξή σημείο, αν κατάλαβα αυτό που ρωτήσατε, ο κ. Καρκόφ μόλις ανέφερε, Δηλαδή όχι μόνο να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο οργανισμό πέρα από την Frontex, την Europol, τη CITSEN, οι άλλες, δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα έργα που πρέπει να επιτελεστούν. Χρειάζεται επαγγελματισμός και να τα ανακατέψετε όλα μαζί. Νομίζω ότι ίσως ε, αυτή η μέθοδος δεν θα είναι η πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό θα ήμουν προσεκτικός προτού προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Η τελευταία παρατήρηση είναι, έχει σχέση η σχέση με το θέμα των παραδόσεων. Εάν θυμάμαι καλά, πώς μπορούμε να το πούμε. Αυτές ήταν προσπάθειες από την κυβέρνηση Μπούς να πείσουν όχι όλα τα κράτη-μέλη, αλλά μερικά εξ αυτών, να αρχίσουν μια συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που θα παρουσίαζε μια συνεργασία όσον αφορά τις παραδόσεις, οι ενέργειες αυτής της μορφής. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, από ό,τι θυμάμαι, αυτό δεν προχώρησε πολύ, διότι πολλά κράτη-μέλη είχαν μεγάλες δυσκολίες να προχωρήσουν με αυτή την πρόταση. Για τον απλούστατο λόγο ότι πολύ συχνά ε, μπορεί κανεί να ε, παραβιάσει θεμελιώδεις αρχές ε, του δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Γι' αυτό ε, όταν άλλαξε η κυβέρνηση και ήρθε ο Ομπάμα δεν προχώρησε αυτή η ιδέα διότι η κυβέρνηση Ομπάμα η ίδια δεν ήθελε να προωθήσει αυτό το θέμα διότι ήδη έχει δυσκολίες με το θέμα του Γκουαντάναμο και πώς μπορεί να βρει μια έξοδο από αυτό το σύστημα και νομίζω, <laughs> φυσικά δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω δεν συζητήθηκε περαιτέρω αυτό το θέμα όπως γινόταν με την προηγούμενη κυβέρνηση της Αμερικής. Αυτά ήθελα να προσθέσω. Ευχαριστώ. We thank you both Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Κύριε σάλμι και Δημό, ο κύριο Σάλμη θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, εντάχει, ως προ θέματα που εφήγησαν και ίσω δεν απάντησα ακόμα. Σε επίπεδο ε, αντιμετώπισης τρομοκρατίας ερωτήθηκα κατά πόσο έχουμε προβεί σε ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δηλαδή, κατά πόσο είμαστε μία μονάδα αντιτρομοκρατίας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν θέματα ασφάλειας κάργο και αεροπλοείας όπου ε, συνεισφέρουμε και εμείς για λήψη πολιτικών αποφάσεων, αλλά όχι σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Βημό, ο αντιπρόεδρος ΕΙΕΘ και ο κύριος Σάλμι, ο διευθυντής της ΣΥΤΤΣΕΝ. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να υποβάλλετε και άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Μισελ, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Προς τον κύριο Βημό. Δέχομαι την προσέγγιση και θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Βημό, αφού άκουσα όλες αυτές τις επεξηγήσεις, θα ήθελα να μάθω το εξής. Τι λείπει από την AEDF, ε, ε, ε, ποιες είναι οι ελλείψεις δηλαδή σε σχέση με το υπάρχουν και μη υπάρχουν. Έχετε το λόγο κι εσείς. Ευχαριστώ δύο ερωτήσεις. Πώς αντιμετωπίσετε το θέμα της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο και πώς μπορείτε να αναλύσετε τα, τα δεδομένα Mrs. Entveld, another point. Των Black Swans, των μαύρων κύκνων, ρώτησε ο μιλητής. Κυρία όπως είπε και ο Γιάννα Άλμπρεχτ, ε, υπάρχουν ε, ε, θέματα δημοκρατικού ελέγχου, κοινοβουλευτικού ελέγχου, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει το Εθνικό Κοινοβούλιο στα κράτη-μέλη. Εσείς ε, σε τι κοινοβουλευτικό έλεγχο υπόκειστε, σε ποιον είστε υπόλογοι, αν δεν είστε υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα ξανανοίξουν τη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία ερώτηση, ο κ. Σάριος Βόλσκι. Ο κ. Σάριος Βόλσκι πρώτα και άλλος ένας ομιλητής το ΣΥΤΣΕΝ ακούσαμε ότι δεν ε, συλλέγει πληροφορίες, δεν είναι υπηρεσία πληροφοριών. Χρειαζόμαστε ε, ένα κοινό σύστημα συλλογής πληροφοριών, όπως προτείνουν ορισμένοι συνάδελφοι και με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας εβδομάδας. μέρα και Ρομπέρτο Έχω ορισμένες αμφιβολίες σε σχέση με την ε, κατάφαση ότι η συνθήκη δεν θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει πληροφορίες, να έχει μια δική της υπηρεσία. Γιατί θα πρέπει να βασιστούμε σε πληροφορίες από άλλους φορείς. Δίας μέρα, παρακαλώ, σύντομα. Ευχαριστώ τηλεγραφικά, επειδή έφτασα αργά. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς ενδεχόμενες αμφιβολίες που υπάρχουν. Υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών, με έχουμε το Frontex, την Europol, την Eurojust και στον αντίποδα έχουμε τον συντονιστή κατά πολέμηση της τρομοκρατίας και τον επόπτη προσωπικών δεδομένων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές κατά πόσο αυτά αυτά τα, αυτοί οι φορείς έχουν επιχειρησιακή δραστηριότητα, μα μόνο η Frontex έχει επιχειρησιακή δραστηριότητα. Άρα όταν μιλάμε για κοινοβουλευτικό έλεγχο, για ποιο έλεγχο μιλάμε τη στιγμή που λαμβάνονται πληροφορίες, υπάρχει intelligence, πώς προωθείται. Θα πρέπει αυτό να καταστεί απόλυτα σαφές. Θα πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος ως προς ε, φορείς ασφάλειας που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία, γιατί διαφορετικά κάνουμε ένα copy-paste πληροφοριών. Θα ήθελα αυτή τη ε, διευκρίνηση και από την άλλη πλευρά της στάθμης να δούμε κατά πόσο έχουμε ένα φορέα ελέγχου που είναι ο επόπτης καθώς και η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Βημό, τελικός γύρος απαντήσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη φορά θα μιλήσω γαλλικά για να αλλάξουμε λίγο και για να απαντήσω και προς τον κύριο Υπουργό. Και βέβαια, δεν θα μπορούσα να πω και τίποτα άλλο εξάλλου, που έχω το συνάδελφο δίπλα μου. Και βέβαια είναι χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να το εφεύρουμε και εξάλλου το εφήβραμε διότι ε, το Συμβούλιο θεώρησε σκόπιμο μετά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση ε, να υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση ε, που θα χρησιμοποιεί όλε τι ανοιχτέ πηγέ. Θέλουμε να έχουμε μια σύνθεση όλων των ανοιχτών πηγών, κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε εύκολο και μας δίνει ένα τελικό προϊόν πάρα πολύ χρήσιμο. Καθημερινά, πολλές φορές κάθε μέρα μας είναι χρήσιμο γιατί καθημερινά το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων μας δίνει πληροφορίες πολύ χρήσιμες. Και επίσης έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που δίνουν τα κράτη-μέλη, των οποίων τη σύνθεση εξασφαλίζει το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων. Αυτές είναι υπηρεσίες πάρα πολύ χρήσιμες και το ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες δεν μας εμποδίζει να θα σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση των δεδομένων τη σύνθεση των πληροφοριών που κάνει το κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Θα προχωρούσαμε στα τυφλά χωρίς αυτή την ανάλυση που κάνει το ΣΥΤΣΕΝ. Είναι λοιπόν πραγματικό πλεονέκτημα και πραγματικά προσθέτει αξία το κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Δεν φαντάζομαι ότι περιμένετε να σας πω και τίποτα άλλο, αλλά πραγματικά αυτή είναι η ειλικρινή μου άποψη. Όσον αφορά το θέμα του πολιτικού ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, από την οποία εξαρτάται το κοινό κέντρο επιχειρήσεων, όπως επίσης και η Στατιωτική Επιτροπή και άλλες υπηρεσίες. Είναι μια υπηρεσία υπό το δικό σας έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι υπό τον έλεγχο βάση, τον έλεγχό σας βάσει των διατάξεων της συνθήκης και άλλων κανονισμών. Ο πολιτικός έλεγχος λοιπόν υπάρχει, όπως και για τη Frontex, που εξαρτάται από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, ο ίδιος έλεγχος μπορεί να υπάρχει μέσω των επιτρόπων δεν θα πρέπει να συγχαίουμε δύο θέματα. Το γενικό πολιτικό έλεγχο που υπάρχει μέσω των πολιτικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΥΠΑ εκπροσώπου αφενός και το θέμα των εγγράφων ε, εμπιστευτικού ή απολύτου χαρακτήρα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα έγγραφα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα τα οποία δεν, δεν πρέπει να συγχαίουμε. Η πρόσβαση στα εμπιστευτικά έγγραφα είναι κάτι το διαφορετικό. Ήδη έχουμε κάποιους κανόνες και θεσπίζουμε συγκεκριμένες διατάξεις και πρέπει να γίνει σαφώς η διάκριση μεταξύ των δύο. Ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο μας θέσατε και πάλι ήταν γιατί δεν θα ήταν σκόπιμο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, ένα ευρωπαϊκό οργανισμό πληροφοριών και ασφάλειας που θα μπορούσε να έχει δικές του δραστηριότητες, δικές του πληροφορίες. Κύριε Σάριος Βόλσκι, θα σας απαντούσα ότι είναι κάτι που μοιάζει με την εξωτερική πολιτική. Βρισκόμαστε σε μια κοινή εξωτερική πολιτική, δεν έχουμε μια ενιαία εξωτερική πολιτική. Ίσως κάποια στιγμή να φτάσουμε και σε αυτό το στάδιο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Το να θέλουμε να βάλουμε πάνω από όλες τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών μια ευρωπαϊκή πληροφορία θα δημιουργούσε επικάλυψη, κατά τη γνώμη μου, που θα ήταν εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών της Ευρώπης. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε μια τέτοια πορεία πρέπει να κάνουμε συνετά βήματα με την προοδευτική, με την ε, συμφωνία των κρατών μελών σιγά σιγά. Έχουμε κάνει ήδη αρκετά βήματα και έχουμε επιτύχει προς το παρόν μια σημαντική πρόοδο και ο Ήλκα ο πρόεδρος του ΣΥΤΣΕΝ θα μπορούσε να σας πει πολύ περισσότερα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών δέχτηκαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να θέτουν τις πληροφορίες τους ε, ε, από κοινού και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν από χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημό και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ήλκα Σάλμη και πάλι εκ μέρους του Κοινού Κέντρου Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος γιατί δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε ο κύριος Βημό για το αν είμαστε υπόλογοι σε κάποιο εθνικό κοινοβούλιο, η απάντηση είναι όχι, δεν είμαστε υπόλογοι σε κάποιο εθνικό κοινοβούλιο. Ίσως ε, ε, κάποια άλλη φορά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τα θέματα πηγών πληροφοριών ε, που έχουμε. Αυτά προ το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε και του δύο, και τον κύριο Σάλμη και τον κύριο Βημό. Και ευχαριστούμε και τα μέλη τη Επιτροπή ΣΕΝΤΑ και τη Επιτροπή ΑΦΕΤ που ήρθαν σε αυτή την κοινή συζήτηση. Και περνάμε στο επόμενο σημείο τη μερίσια διάταξη, ε, αποχαιρετώντα του προσκεκλημένου μα. We thank. We thank Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΣΑΦΕΤ και της Επιτροπής City. Παρακαλώ ησυχία, καθώς φεύγετε. Thank you, colleagues, συνάδελφοι, θα ήθελα την προσοχή σας για να περάσουμε στο σημείο 5 που αφορά τη συνολική προσέγγιση ε, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, αυτό το σημαντικό φάκελο, για το οποίο θα αφιερώσουμε 30 λεπτά. 30 λεπτά για να ακούσουμε την παρουσίαση ε, του σχεδίου εισήγηση και την ανακοίνωση της Επιτροπής. Ο συνάδελφός μας, ο κύριος Άξελ Βος, είναι εισηγητής επί του θέματος. Θα μας μιλήσει ο εισηγητής, θα παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδίου έκθεσης και μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση για να μιλήσουν οι συνάδελφοι που το επιθυμούν. Θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για την ε, κατάθεση των τροπολογιών είναι 26 Απριλίου το μεσημέρι. Κύριε Φως, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεση σχετικά με τη συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχω παρουσιάσει το έγγραφο εργασία και γι' αυτό σήμερα θα είμαι πολύ σύντομο ε, να σα πω ποιο είναι το γενικό πλαίσιο για, την έκθεση, για το σχέδιο έκθεση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ε, μια οδηγία ορόσημο ε, για ε, τα θέματα προστασίας των δεδομένων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 15 χρόνια αρχίσαμε να έχουμε αυτές τις διατάξεις και στο μεταξύ η τεχνολογία έχει προωθήσει όπως επίσης και η νομική κατάσταση μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει τροποποιηθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να προσαρμοστεί η οδηγία δεν εφαρμόζεται παντού ομοιόμορφα και στον τομέα ε, του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ε, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διατάξεις. Ε, περιμέναμε μια ανακοίνωση της Επιτροπής τον Ιούλιο πριν από, την, από τις καλοκαιρινές διακοπές και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξουμε πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι μπορούσαμε να παίξουμε το 1995 είναι ένα καθήκον το οποίο αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα και γι' αυτό χαίρομαι για τη δυνατότητα που θα έχουμε με αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας να δηλώσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μαζί με το Σκιώδη Συγητή διαμορφώσαμε αυτό το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τα βασικά θέματα που ενδιαφέρουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, λόγω των περιορισμών της έκθεσης πρωτοβουλίας δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε λεπτομερώς διάφορα θέματα. Προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στα βασικά και σημαντικά θέματα και ε, υπάρχουν πέντε βασικά σημεία τα οποία προτείνουμε. Καταρχήν, πλήρη ε, εναρμόνιση των υφισταμένων ε, κανόνων για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου σε αυτό το τομέα. Δεύτερον, επέκταση της προστασίας και στους τομείς δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Τρίτον, διευκρίνηση των κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό τόπο ενός διαμετακομιστή ή του υπευθύνου φορέα προστασίας δεδομένων, για να έχουμε ίδιο επίπεδο προστασίας των ατόμων. Τέταρτο σημείο, ενδυνάμωση των δικαιωμάτων ε, ε, του ατόμου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τον έλεγχο των δεδομένων αυτών και πέμπτον αποτελεσματική εφαρμογή ε, και ευθυγράμμιση των διατάξεων για την προστασία δεδομένων. Αυτά είναι επιγραμματικά τα βασικά σημεία για το ε, σύστημα προστασίας των δεδομένων. Μας ενδιαφέρουν και οι δυνατότητες αυτορύθμισης που μπορούν να υπάρχουν για να συνοδεύουν αυτές τις βασικές διατάξεις. Το θέμα της προστασίας των δεδομένων δεν είναι ένα θέμα το οποίο το εφήβραμε τώρα ή που μας προέκυψε τώρα. Έχουμε ήδη μία οδηγία από το 1995, όπως σας είπα, ε, που τώρα πλέον ε, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί για να καλύπτει τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Με χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας ε, και θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου πριν ανοίξει η συζήτηση. Θα ήθελε κάποιος εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος της ε, Προεδρίας να λάβει το λόγο ή εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς από πλευράς Επιτροπής ε, επιδεικνύουμε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση που υποστηρίζει τις προτάσεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής και περιμένουμε την άποψη του Κοινοβουλίου επί του θέματος με βάση το νομικό μέσον που θα παρουσιάσει η Επιτροπή μετά το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Το Συμβούλιο, η Προεδρία θα ήθελε να κάνει μια ανακοίνωση, μια εισήγηση, φαίνεται πως όχι. Άρα ξεκινάει η συζήτηση και αρχίζουμε την κυρία Ιντβέλτ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω το σχέδιο γνώμης του εισηγητή, ο οποίος συνεργάστηκε με τους σκιώδεις στενά, άρα δεν μας εξέπληξε το αποτέλεσμα. Υπάρχουν ορισμένα, ορισμένες βασικές αρχές στην έκθεση. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο πρώτο τύπο προστασίας προσωπικών δεδομένων και βεβαίως ε, για ειδικού τομεί θα υπάρξουν ειδικέ διευθετήσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα νέο μέσο που να καλύπτει και τον παλαιό πρώτο πυλώνα και τον ίν τρίτο. Ως προς την εναρμόνιση, νομίζω ότι υπάρχει επαρκής ε, συνένεση για εναρμόνιση, που ενδιαφέρει και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, διότι το σύστημα θα έχει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα ήταν σκοπιμότερο να χρησιμοποιήσουμε κανονισμό και όχι οδηγία στο μέτρο του δυνατού. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο αποτελεί και πρόκληση είναι η παγκόσμια διάσταση γιατί μπορούμε ενδοκινοτικώς να συντονιστούμε αλλά δεν μπορούμε να περιορίσουμε τα δεδομένα που ε, διατίθενται ανά τον κόσμο. Δεν περιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Παρατήρησα από τον τύπο την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Αυστραλία προβάλλει ένα νέο σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων με πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας για τους πολίτες της και ως προς το θέμα της ε, θέσης σε ισχύ, νομίζω ότι το θέμα της λογοδοσίας που έχουν καταρτήσει πολλά εμπλεκόμενα μέρη είναι ένα κέριο θέμα. γιατί η θέση σε ισχύ της ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αφορά ε, απλώς ε, μία, το ότι σταυρώνουμε συγκεκριμένα τετραγωνίδια. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Είναι κάτι ένα θέμα ύψης της σημασίας. Θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση κατάχρησης προσωπικών δεδομένων, διότι έχουν γίνει τόσο σημαντικά στην ε, καθημερινή μας ζωή τα προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε αν υπάρχει κατάχρηση να υπάρχουν και σοβαρές κυρώσεις. κυρία Ζίμπελ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που για άλλη μια φορά ασχολείται με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν ουσιαστικά θέματα σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα οποία μας τόνισε ο συντονιστής. Ιδίως στο σημείο 8 της έκθεσης για την καμπάνια ευαισθητοποίησης, βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό. Σε κάθε τομέα της ζωής, στον τομέα της αναψυχής, στον επαγγελματικό τομέα, στον οικονομικό τομέα, στον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων, υπάρχουν αυτά τα θέματα και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδίως οι νέοι να ενημερώνονται Ξέρουμε ότι οι νέοι χρησιμοποιούν τα νέα μέσα με μεγάλη ικανότητα, αλλά δεν έχουν επίγνωση των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν όταν δίνουν προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, όταν κάνουν αγορές από το διαδίκτυο κλπ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πιστεύω ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και να υπάρξει και υλικό για την κατάρτιση των νέων και για να βελτιωθεί η ικανότητα των νέων να χειρίζονται το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σάλβαρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Φαίνεται ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να τονίσει τη σημασία της προστασίας δεδομένων Θα ήθελα να πω κάτι ως υποσημείωση. Η πρόταση της Επιτροπής, μας είπε η Επιτροπή ότι θα υποβληθεί μετά τις διακοπές, ενώ εγώ, μετά τις διακοπές. Εγώ περίμενα ότι θα υποβληθεί η πρόταση της Επιτροπής πριν από τις διακοπές. Κύριε συνάδελφε, κύριε Φως, πρέπει να τολμήσουμε και να ζητήσουμε κανονισμό και όχι οδηγία γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη να το κάνουν όπως θέλουν. Είτε θέλουμε εναρμόνιση, οπότε θα περιμένουμε να έχουμε κανονισμό και θα ε, υποστηρίξουμε και την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ για να έχουμε τελικά κανονισμό. Γιατί αν πούμε ότι ε, θέλουμε να έχουμε κάποια εναρμόνιση, δεν θα μας οδηγήσει στην επιθυμητή εναρμόνιση. Η ευαισθητοποίηση ε, είναι πολύ καλή ιδέα και μπορεί να είναι κάτι το οποίο ως συνοδευτικό μέσο θα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί θέλουμε ε, να έχουμε πολίτες οι, οποίες, ε, οι οποίοι ε, από μόνοι τους μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις για το πώς θα χειριστούν το θέμα της παροχής δεδομένων στο διαδίκτυο. Και όταν δίνουν δεδομένα σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και όταν κάνουν αγορές στο διαδίκτυο και για διαφημίσεις. Είναι σημαντικό να είναι εκπαιδευμένοι οι πολίτες ώστε να μπορούν να έχουν την απαραίτητη ελευθερία απόφασης. αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε είναι αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τα δεδομένα να είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν ποια θα είναι η χρήση των δεδομένων την οποία θα κάνουν. Και από αυτό το οποίο έγινε στην Αυστραλία νομίζω ότι μπορούμε να διδαχτούμε θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα πιστοποιητικό για την χρήση των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσουμε το θέμα της εδαφικότητας. Θα μπορούσαμε να έχουμε προτυποποίηση όπως το ISO 2009 ε, για να έχουμε ένα είδος πιστοποίησης ε, για, ε, τα δεδομένα, για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα από το που προέρχονται, αν προέρχονται από το Μπακού ή από την Βόνη. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάτι τέτοιο για να μπορούμε να έχουμε σωστή προστασία των δεδομένων. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσε να πει κανεί, δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ελπίζω να προκύψει κανονισμό από αυτή την πρόταση και να έχουμε τον χρόνο να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ένστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θετικό είναι ότι ε, ζητάμε την εναρμόνιση και μάλιστα σε όλους τους τομείς. Είναι κάτι το οποίο ε, συγκρούεται με την πολιτική της κυβέρνησής μας σχετικά με, το, με τη χρήση των πληροφοριών στον, στον τομέα αστυνομική και δικαστική ε, συνεργασία. Εμένα με ενδιαφέρει το ποια είναι η άποψη του εισηγητού ε, σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων και την προστασία τους ε, σε αυτό το τομέα. Ήταν ενδιαφέρουσα και η άποψη ότι πρέπει να έχουμε ένα κανονισμό και όχι οδηγία για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική εναρμόνιση. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ένα δεύτερο σημείο σχετικά με τις τρίτες χώρες υπάρχει μια ήπια διατύπωση σχετικά με τις τρίτες χώρες και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερέστερα για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Το θέμα του επόπτη προστασίας δεδομένων και οι δυνατότητες ελέγχου και οι αρμοδιότητες είναι πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο Συμβούλιο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια διατύπωση ακριβέστερη σε αυτό το σημείο και στην, ε, στο έγγραφο της Επιτροπής να υπάρξει μια διατύπωση ε, ακριβέστερη. Για το θέμα των κυρώσεων που μίλησε η κυρία Ιντβελντ ε, και εγώ το είχα εντοπίσει αυτό το θέμα, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περαιτέρω. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η συνεργασία με τον κύριο Φως, τον εισηγητή, ε, είναι πολύ καλή και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την έκθεσή μας. Η έκθεσή μας μιλά για την ανακοίνωση της Επιτροπής από το πέρυσι το φθινόμπορο ε, και ε, είναι σημαντικό να πούμε ότι η οδηγία 9546 για μας είναι η αφετηρία για την μεταρρύθμιση που απαιτείται. και είναι σημαντικά αυτά που είπε και ο εισηγητής για να δούμε αν θα προχωρήσουμε ε, σε μια οδηγία ή σε ένα κανονισμό. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να έχουμε ένα κανονισμό αλλά σίγουρα δεν ε, αμφισβητούνται αυτά τα οποία έχουμε πει για την προστασία των δεδομένων. Και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε συμπεριλάβει και το θέμα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 16 προστατεύεται και η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. είναι σημαντικό όταν θα συζητάμε την οδηγία ή τον κανονισμό, αυτό το οποίο θα μας απασχολεί να είναι η καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές δυσκολίες, ιδίως στις εξωτερικές σχέσεις, στη συμφωνία ΣΕΦΑ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, και ελπίζω ότι θα υπάρξει καλύτερη διασφάλιση στο μέλλον. Ευχαριστώ. κύριε Ρωμέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή το εξής. Επειδή εκφράζεται γενικά, με γενικούς όρους, πώς η προστασία δεδομένων μπορεί να ενταχθεί σε μια διεθνή συμφωνία γιατί αυτή είναι η βάση των δικών μας προδιαγραφών που θα πρέπει να, να υπερασπιστούμε έναντι των ΙΠΑ, ας πούμε, δηλαδή σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που γίνεται με τις ΣΥΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας. Εάν η οδηγία ε, ξεπερνιέται από την ε, νομολογία των κρατών μελών ή αν έχει ενταχθεί ή όχι στις εθνικές ένομες τάξεις, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Εν πάση περιπτώσει, οι γενικές ενιές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και με άλλα κράτη. Γιατί αν δεν έχουμε μία συνεκτική νομοθεσία θα είναι δύσκολο να απαιτήσουμε κάτι τέτοιο από άλλα κράτη. Και εδώ μιλώ ιδιαίτερα για τις διαπραγματεύσεις τι τον είπα. Ο κύριος Μπρόγκς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πρόβλημα με την ουσία του μεγαλύτερου μέρου έκθεση. παρά το γεγονό. ότι θα προτιμούσα να πούμε ότι είναι ε, μια διεθνή συμφωνία παρά ένας ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ας το αφήσουμε κατά μέρος. Αν όμως ε, δούμε το σημείο Δέλτα συγκεκριμένα, λέμε ότι αυτό είναι ένας κίνδυνος προφάλι ναι, όταν υπάρχουν ε, μεγάλα εγκλήματα, κυρίως η τρομοκρατία. Το προφίλ είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει κανείς καλά, θεωρείται ότι συνιστά διάκριση. Όταν πρόκειται όμως ε, να βρούμε υπόπτους, τότε είναι φυσιολογικό να κάνουμε έρευνες ε, για τα άτομα τα οποία έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα όσον αφορά το προφίλ. Ο κύριος Φως, μετά τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ελπίζω να μπορέσω κάπως ε, να ρίξω λίγο φως στο σκοτάδι. Ε, καταρχήν σε σχέση με αυτό που αναφέρεται για την Αυστραλία δεν το γνωρίζω καθόλου το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξή σας. Θα μπορούσαμε και διμερώς να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ο Αλεξάνδρ έφυγε. Όσον αφορά τον κανονισμό, νομίζω ότι είναι διτή η προσέγγιση. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία το μέσο που θα επιλέξουμε όσο το περιεχόμενο το οποίο θα επιλέξουμε και θα πρέπει ε, ε, ε, να φροντίσουμε την ποιότητα του περιεχομένου. Αν έχουμε ένα χαλαρό κανονισμό ή μια αυστηρή οδηγία μπορούμε να επιτύχουμε νομίζω το σκοπό μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν μιλάμε για εναρμόνιση, όμως μάλλον κινούμεθα προς την κατεύθυνση του κανονισμού. Ε, νομίζω ότι ε, από τις συζητήσεις μας ε, αυτά τα οποία προέκυψαν με οδήγησαν σε αυτά τα οποία έχω συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσης. Ε, προς την κυρία Ένστ όσον αφορά την εναρμόνιση και τη σύγκρουση με τις πολιτικές εθνικών κυβερνήσεων θα ήθελα να πω ότι για μένα αυτό που έχει προτεραιότητα είναι καταρχήν να έχουμε ένα λογικό σύστημα προστασίας των δεδομένων ε, και θέλουμε να δούμε πώς θέλουμε να προστατεύεται ο πολίτης είναι δευτερεύουσα σημασία να δούμε το τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Εμεί αυτό το οποίο πρέπει να προωθήσουμε είναι ένα λογικό σύστημα για το οποίο εμεί θα θεωρούμε ότι παρέχει λογική, επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό πρέπει να είναι το σενάριο από το οποίο θα ξεκινήσουμε. Όσον αφορά τον επόπτη προστασίας δεδομένων ε, ή της ε, μαζικές ε, αγωγές. Ε, δεν αρκεί αυτό το έγγραφο. Έχουμε ζητήσει ε, κάποια θέματα και θα χρειαστεί να κάνουμε και κάποιες τροποποίησεις και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε τις γενικές γραμμές πάνω στις οποίες θα τονίσουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα σημαντικά θέματα για μας. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες μπορούμε να τις συζητήσουμε όταν θα περάσουμε σε πιο λεπτομερή εξέταση των θεμάτων. Προς την κυρία Ρομέρα και τον κύριο Μπρόνς ε, σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες που αναφέρατε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο κάνουμε εμείς για μας τους ίδιους και για τους πολίτες μας. Οι διεθνείς ε, συμφωνίες ε, θα ακολουθήσουν. Εμείς μπορούμε να θέσουμε τα πρότυπα για αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε λογικό και απαραίτητο και αυτό το οποίο θα θεωρούμε και λογικό για τις διεθνείς συμφωνίες. Αυτό το οποίο έχουμε ήδη στην οδηγία είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε ως αφετηρία και μπορούμε από ε, αυτού να προσαυξήσουμε αυτά τα οποία θα θελήσουμε να έχουμε από τις διεθνείς συμφωνίες. Ε, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις καθώς και αποζημιώσεις ε, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε και στο διεθνή τομέα προς τον κύριο Μπρόντς για το σημείο Δέλτα που αναφέρατε για το profiling, τη διαμόρφωση εικόνας προσώπου. Αυτό δεν αφορά τις κρατικές αρχές αλλά οι τεχνικές δυνατότητες ε, αυτή τη στιγμή έχουν προδεύσει τόσο πολύ που είναι πολύ εύκολο ε, σε ηλεκτρονικό περιβάλλον να διαμορφωθεί το προφίλ, εικόνα, του προσώπου, εικόνα προσώπου ενός ατόμου. Γι' αυτό μιλάμε για κίνδυνο του, της διαμόρφωσης εικόνας προσώπου σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή η εικόνα η οποία διαμορφώνεται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φως. Ε, εάν θέλετε να θίξετε ένα θέμα, θίξτε το εντάχει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γρήγορα. Χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βος, διότι η έκθεση είναι εξαιρετική. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για ενίσχυση εθνικών εγγυήσεων και παράλληλα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το άρθρο 29 το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και ίσως η ομάδα αυτή θα πρέπει να μετατραπεί σε υπηρεσία, σε αυτόνομη υπηρεσία. Έγινε λόγος για profiling, ότι απαγορεύονται αυτές οι δραστηριότητες profiling και ίσως θα μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες για πολίτες αλλά τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα χειριστούν μόνο ε, φορείς και υπηρεσίες αρμόδιες. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά την ενίσχυση των εθνικών εποπτών προστασίας δεδομένων, ένα θέμα που ανέφερε και η κυρία Έρνστ, όπως επίσης και όσον αφορά την ομάδα εργασίας 29 του άρθρου 29. Με βάση τις προτάσεις που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορέσουμε να δούμε πολύ συγκεκριμένα πώς μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι δηλαδή απομονωμένα για συγκεκριμένα σημεία, αλλά ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα, θα μπορέσουμε να το έχουμε και να καλύπτει όλους τους τομείς χωρίς κενά κάτι το οποίο θα έχει εφαρμογή και για τους Εθνικούς Επόπτες Προστασίας Δεδομένων και για την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Δεν θέλουμε να υπάρχουν παράλληλες εργασίες, αλλά να υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή κατά νουν. Όσον αφορά την απαγόρευση του profiling, το έχουμε συζητήσει εδώ το έχουμε συμπεριλάβει πολύ περιληπτικά, δεν είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε λεπτομέρειες. Ενδεχομένως ε, μπορούμε να υποβάλουμε μια κοινή τροπολογία για το θέμα αυτό και για τις ε, πληροφορίες ε, και για το δικαίωμα προστασίας. Νομίζω ότι είναι ε, κάτι για το οποίο υπάρχει συμφωνία με το σκιώδη εισηγητή. και ήδη η βάση υπάρχει στην οδηγία του 95. Πάντως ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και να προχωρήσουμε επί του θέματος. Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε κύριε Φως, λέει ο Πρόεδρος. Είδαμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης και αποφασίσαμε για τις προθεσμίες για την κατάθεση των τροπολογιών. Και το επενθυμίζω, 26 Απριλίου μέχρι το μεσημέρι. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο σημείο 6, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Δηλαδή πολιτική αντιτρομοκρατίας ε, της ε, Ευρώπης, βασικές ε, επιτεύξεις και μελλοντικές προκλήσεις. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 6. Όπως είπαμε, αφορά το σχέδιο έκθεσης της συναδέλφου κυρίας Εντβέλτ όσον αφορά την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, αντιτρομοκρατίας και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια ακρόαση του θέματος Τώρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια να μας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του σχεδίου έκθεσης και κατόπιν θα ανοίξω τη συζήτηση ώστε να κάνετε τα σχόλιά σας καθώς και ε, την Επιτροπή και το Συμβούλιο αν θέλουν να παρέμβουν. Σας υπενθυμίζω ότι όπως και στην προηγούμενη περίπτωση η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 26 Απριλίου το μεσημέρι. Κυρία Συγκήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι αρκετά σύντομη, επειδή ήδη είχε γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με βάση το αρχικό έγγραφο εργασία μου. Αυτό που έχετε μπροστά σας τώρα είναι η σύνοψη των εγγράφων εργασία. Δεν έχω κάνει αλλαγές απλά και μόνον. Είναι πιο βραχή το κείμενο. Και υπάρχουν και οι επειδή υπάρχει περιορισμένο αριθμό σελίδων που μπορούν να μεταφραστούν και δεδομένου ότι ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες εξαιρετικέ προτάσεις από τους συναδέλφους, σας παροτρύνω να καταθέσετε τροπολογίες αν θέλετε. Όσον αφορά στη διαδικασία τώρα, ορισμένες πρακτικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όταν γίνεται, να απαντήσουν ήδη στα ερωτήματα που τέθηκαν στην έκθεση. Τίποτα δεν τους αποτρέπει να το κάνουν. Και ορισμένα από τα ερωτήματα είναι αρκετά σαφή. Δηλαδή, ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή ε, ποιες γραμμές του προπολογισμού αφορούν την αντιτρομοκρατία. Αυτή τη στιγμή ή μάλλον έχει ήδη ανατεθεί μία ε, μελέτη από την Επιτροπή μας και θα έχουμε ε, τα αποτελέσματα στο τέλος του μήνα και τα προκαταρτικά αποτελέσματα πριν από την ακρόαση στις ερχομένες εβδομάδες για να έχουμε μια γενική ιδέα και τελικά είναι δύσκολο να δούμε πόσα χρήματα ξοδεύουμε για την αντιτρομοκρατία. Η Επιτροπή κάθε χρόνο παρουσιάζει τον ετήσιο προπολισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση Έχετε τους ανθρώπους που γνωρίζουν σίγουρα, που γνωρίζουν πόσα χρήματα ε, προβλέπουν για την αντιτρομοκρατία. Πέρσι ο αξιωματούχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μίλησε είπε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, με συγχωρείτε, γιατί είναι πολύ φιλόδοξη αυτό το σχέδιο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Επί τη ουσία τώρα. Ή μάλλον, μία τελευταία παρατήρηση επί τη αρχή. Γιατί, γιατί γίνεται αυτή η άσκηση. Όχι επειδή δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε μια αντιτρομοκρατική πολιτική, πολιτικές που θα είναι αποτελεσματικές και που θα έχουν και νομιμότητα δημοκρατική. Γι' αυτό είναι αξιοθαύματο το γεγονός ότι ε, έχουμε χαράξει εδώ και 10 χρόνια αυτές τις πολιτικές αντιτρομοκρατίες χωρίς να ξέρουμε Πού καταλήγουμε. Νομίζω ότι ο κύριο Μπρόγκ το έθιξε αυτό το θέμα με πολύ ζωντανό τρόπο στη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, αυτές οι αντιτροποκρατικέ πολιτικές των 10 ετών τι πέτυχαν. Δεν το γνωρίζουμε. Πόσο κοστίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Ποιε είναι οι επιπτώσεις ε, στις πολιτικές ελευθερίες. Δεν το γνωρίζουμε. Ποτέ δεν μετρήθηκαν, ποτέ δεν αξιολογήθηκαν δεν υπάρχει άλλο τομέα πολιτική που να μην υπόκειται σε δημοκρατική αξιολόγηση και έλεγχο Εκτό από αυτόν τον τομέα. Είδα ορισμένα πρώτα αποτελέσματα τη μελέτη, την οποία μόλι ανέφερα, όσον αφορά τι οικονομικέ πλευρέ. Υπάρχει μεγάλο κατάλογος μέτρων που προτάθηκαν από την Επιτροπή και υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι από τον κατάλογο, αυτό το μεγάλο κατάλογο, μόνο δύο ε, ήταν αντικείμενο εκτίμηση των επιπτώσεων. Νομίζω ότι πουθενά αλλού δεν βλέπουμε ένα τόσο μικρό κατάλογο. Νομίζω λοιπόν πάλι καταλήγοντας ότι είναι ουσιαστικό να αξιολογούμε τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές και ορισμένοι θα σκεφτούν ότι αυτό σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι με τις πολιτικές αυτές καθόλου, αλλά θέλουμε οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές να είναι αποτελεσματικές, να καταλήγουν σε αποτελέσματα, να κάνουν αυτό το οποίο υποτίθεται θα κάνουν, δηλαδή να προστατεύουν τη δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή ώστε να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης για να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες πολιτικές. Ευχαριστώ. Ήταν ε, συνοπτική η παρουσίασή σας ενός περίπλοκου ε, και επίκαιρου θέματος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκπροσωπείται η Επιτροπή εδώ από τον κύριο Μάρτιν Σίφερ, ο οποίος θέλει ίσως να μιλήσει. Η Επιτροπή θέλει να μιλήσει. Όχι, δεν θέλει. Όχι, δεν είμαι Μάρτιν Σίφερ. Δεν είμαι ο Μάρτιν Σίφερ. Αν θέλετε, παρακαλώ να μας πείτε το όνομά σας. Λοιπόν, ε, sorry, σε την Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων, ο ε, συνάδελφος Μάρτιν Σίφερ θα μιλήσει. Είναι όρθιος. Μόλις έφτασε. Μόλις φτάσατε τη σωστή στιγμή. Την κατάλληλη στιγμή. σας ε, έκαναν ε, μία εισαγωγή ήδη. Αναμένουμε σχόλια της Επιτροπής για την ε, αξιολόγηση της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος και ζητώ συγγνώμη που έφτασα αργά εξετάσαμε το σχέδιο έκθεσης, τα συμπεράσματα και πράγματι ε, πρέπει πολλές δράσεις να ληφθούν για να αξιολογήσουμε όλες τις πλευρές ε, στον τομέα της αντιδρομοκρατίας και αυτό έχει σχέση με τις συζητήσεις που είχαμε σε αυτήν την Επιτροπή στο τέλος Ιανουαρίου με βάση τα έγγραφα εργασίας. Λοιπόν, είδαμε πώς μεταφράστηκαν σε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Δεν καταλήξαμε ακόμα σε οριστικά συμμεράσματα. Και πρέπει να πω ότι έχουν γίνει πολλές προτάσεις. Ορισμένες είναι εφικτές πιστεύουμε και μπορούν να προωθηθούν από την Επιτροπή. Άλλες νομίζω ε, απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών, διότι οι περισσότερες συστάσεις, οι προτάσεις που έχουν γίνει, απευθύνονται στην Επιτροπή. Και ε, για λόγους αρμοδιότητας και πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Γι' αυτό πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτές. Ορισμένες συστάσεις λοιπόν αφορούν τα κράτη-μέλη. Ε, από καθαρά τεχνική άποψη έχουμε ορισμένους δισταγμούς σχετικά με την, το εφικτό ορισμένων μέτρων. Αλλά ακόμα ε, εξετάζουμε εσωτερικά αυτό το θέμα. Τι λέμε λοιπόν, ότι υπάρχουν δύο ή τρεις συστάσεις τις οποίες σίγουρα μπορούμε να υποστηρίξουμε και άλλες τις οποίες ακόμη πρέπει να μελετήσουμε και για τις οποίες θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά δεν θα έχετε όλη την εικόνα για το τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό ξεπερνάει τα πλαίσια ε, των όσων ε, γνωρίζει η Επιτροπή όσον αφορά ε, τις διμερείς διακυβερνητικές σχέσεις της. Αυτά ήθελα να πω σε συντομία. Ευχαριστώ κύριε Σίφερ. Η Προεδρία του Συμβουλίου έχει τίποτα να πει. Θέλει να παρέμβει. Αν όχι, όχι. Πολύ καλά. Τότε αρχίζει η συζήτηση. Ε, θα έδινα το λόγο στην κυρία Λάτφορντ, αλλά δεν είναι εκεί. Α, εδώ είναι, εδώ είναι. Θέλετε να μιλήσετε πρώτοι. Πολύ καλά, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο καθένας φαίνεται να βρίσκεται στο λάθος μέρος σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να πω για αυτή την έκθεση ότι ορθά είπατε ότι υπάρχουν πολλά νομοθετήματα, πολλά χρήματα που έχουν δαπανηθεί και εκείνο που μας χρειάζεται τελικά είναι να δούμε κατά πόσον τα χρήματα που ξοδεύουμε έχουν ε, ε απόκριση έχουν αντίκρισμα, με συγχωρείτε, ε, επί μία δεκαετία ή μάλλον περισσότερο από μία δεκαετία έχουμε αντιτρομοκρατικές πολιτικές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία εσωτερικής ή, ή μη εσωτερικής τρομοκρατίας. Και γι' αυτό κάπως αντιδρούμε όταν οι φίλοι μας πέραν του Ατλαντικού μας λένε ότι δεν ξέρουμε τι λέμε για την τρομοκρατία. Κυρίως όταν ορισμένοι ερετοί στι ΗΠΑ έκαναν πολλά για να χρηματοδοτήσουν και να βοηθήσουν αυτή την τρομοκρατία στο παρελθόν. Υπάρχουν uh, uh, λίγα ερωτήματα. Το ένα είναι το εξής. Ορθά μας λέει η Σοφία ότι όλα τα υπάρχοντα μέτρα θα πρέπει ε, να ε, είναι αντικείμενο ενός τεστ αναλογικότητας. Το θέμα είναι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία να πιστεύουν ότι η τροπολογία του 2008 ε, που ποινικοποιεί την δημόσια πρόκληση τρομοκρατίας στην εσωτερική μας νομοθεσία έχουμε μια τέτοια πρόβλεψη, το κόμμα μου δεν είχε συμφωνήσει, ε, που έχει απαγορεύσει την πρόκληση αν θέλετε. Ε, δηλαδή η ιδέα είναι ότι ποινικοποιείται τα άτομα τα οποία ε, χάρηκαν με τους βομβαρδισμούς του Λονδίνου και της Μαδρίτης και ορισμένοι θεωρούν ότι υπάρχουν επαρκή νομοθετήματα ε, για να κατηγορήσει κανείς αυτούς που έχουν προσπαθήσει να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι απαράδεκτη πρόκληση παρόλο που δεν είναι εγκληματική πράξη. Δεν ξέρω κατά πόσον έχετε παρόμοια εμπειρία αυτής της νομοθεσίας και πόσο φως μπορεί να ρίξει για αυτή τη ροπή να, κάνουμε, να νομοθετούμε συνέχεια. Διότι, ε, αν θέλετε, η τρομοκρατία είναι έγκλημα. Δεν είναι κάτι το, ε, μια διαφορετική δραστηριότητα. Δεύτερον, συζητήσαμε για το profile Είχατε δει ε, ε, κανέναν συνεκτικό ορισμό του profiling της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά αναλύει κανένα τις επιπτώσεις που έχει επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, αν θέλετε, έχω επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό το θέμα η Επιτροπή. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσα να σας μιλήσω για ορισμένα profiling αν ήξερα τι συμβαίνει ακριβώς. Και αν είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις δικλείδες ασφαλείας, στις προστασίες των δεδομένων. Επειδή μπορώ να δεχθώ ε, το, ότι υπάρχει το ψυχολογικό profiling, μπορώ να δεχθώ τη θεωρία ότι το profiling μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην αντιτρομοκρατία, αλλά δεν ξέρω τελικά τι γίνεται. Και δεν ξέρω ποιος το κάνει, εκτός αν δεχτούμε ότι ε, ε, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τα μέτρα ασφαλείας, τις κλίδες ασφαλείας. Και τέλος, η ανακοίνηση Επιτροπής ε, μιλάει πολύ για την αντιριζωστικοποίηση, ένας άλλος όρος και νομίζω ότι είναι ο βίος εξτρεμισμός και όχι η καπικοποίηση. Μετά από πολλά χρόνια στην Επιτροπή ίσως γίνομαι βαρετή. Αλλά κατορθώσατε να βρείτε στοιχεία, δηλαδή όταν υπάρχει το πρόβλημα της χρηματοδότησης ε, της ε, καταστολής, κατασταλτικής αντιτρομοκρατίας, όπως την ονομάζουμε και πώς μπορείτε με χρήματα να βοηθήσετε τις κοινότητες, τις κοινωνίες να καταπολεμήσουν τον εξτρεμισμό. Έχετε βρει τη σωστή ισορροπία. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω και στο ερώτημά μου ότι δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι τις 5.30 έχουμε τρεις προσκεκλημένους σε θέματα ανείχνευσης του, ε, της παρακολούθησης και ανείχνευσης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο θέμα TFTP, η κυρία Χάνκης έχει το λόγο. Ως σκιώδης για αυτή την έκθεση κληρονόμησα αυτή την εργασία εδώ και δέκα μέρες θα μιλήσω ουγγρικά για να μπορέσω να μιλήσω πιο γρήγορα και να είμαι και πιο σαφής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι απόλυτα σαφής. Πρόκειται για μία λογική έκθεση και ιδιαίτερα συνεκτική και συνεπή και να ε, συγχαρώ την εισηγήτρια. Έχω πολλές αμφιβολίες σε σχέση με το ευκταίο, μάλλον με τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της. Υπάρχουν ε, θέματα καθαρά ερευνητικού χαρακτήρα, γιατί από όσο γνωρίζω, ορισμένα θέματα θα ανατεθούν σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή ερευνητές. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο βασικές αξίες. Μιλάμε για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια και είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε μια εξισορρόπηση των δύο πτυχών. Έχω διαβάσει πολλά επί του θέματος από διάφορους ερευνητές και κανένας δεν είναι ανεξάρτητος από τις δικές του ή δικές της αξίες. Και θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς θα επιλέξουμε αυτούς τους εμπειρογνώμονες ερευνητές και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μας εκπροσωπούν σωστά. Ως προς θέμα της επικάλυψης, το σημείο εκκίνησης που είναι σαφές για μένα και που υποστηρίζω είναι ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι απόλυτα ε, σαφές ως προς τα ποσά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Άρα θα πρέπει να αποφύγουμε κάθε μορφή επικάλυψης. Βεβαίως συμφωνώ ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, επικάλυψη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μιλάμε και την ύπαρξη διαφόρων κέντρων. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το Κοινοβούλιο να ξέρει πού και πώς υπάρχουν επικαλύψει. Αυτό, Σόφι, νομίζω ότι αν σκεφτόμαστε σε όρους, ε, με όρους ε, επικουρικότητας, κάτι τέτοιο είναι κοντά στο αδύνατον. Καμία μυστική υπηρεσία δεν θα ήθελε να αποκαλύψει τις εσωτερικές της διεργασίες διότι δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή οποιοδήποτε ε, εργαζόμενου ή πράκτορα για να το πω έτσι. Τώρα, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας είναι δικαιούχος μέτρων καταστολής της τορμοκρατίας, τουλάχιστον στην Ουγγαρία, υπάρχει, υπάρχουν θέμα ε, αλληλένδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά αυτά δεν είναι δημόσια. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να άρουμε αυτά τα προσκόμματα και πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Ως προς το profiling, για τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών, το θέμα αυτό έχει θυγεί πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν μου έχει δοθεί ένας επαρκής ορισμός αυτού του όρου, ιδιαίτερα του profiling της διαμόρφωσης χαρακτηριστικών. Όταν μιλάμε για διαφοροποίηση, για ορισμό της τρομοκρατίας, για προσλήψεις μέσω ίντερνετ, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, δηλαδή και οι δύο ορισμοί του profiling και του data phishing. Ένα άλλο θέμα. Όταν μίλησα με τον κύριο Wainwright, είχα την εντύπωση ότι παλιμπεδίζουμε κάπως, γιατί ζητάμε κάτι, αλλά δεν είμαστε σαφείς για το τι θέλουμε. Τι θέλουμε, γεγονότα, ονόματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις ακριβώς τι εννοείς, χωρίς βεβαίως να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια του οποιοδήποτε. Η αναλογικότητα είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μία δράση καταπολέμησης της τρομοκρατίας ή η αντιτρομοκρατική δράση είναι αναλογική με την απειλή. είναι αντιστρόφως ανάλογη δηλαδή με την απειλή. Θα πρέπει να υπάρχει μία εξισορρόπηση εδώ και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να κρατήσουμε και να στραφούμε στην αρχή της αναλογικότητας. Οι τρομοκράτες μαθαίνουν και πολλές φορές προτρέχουν. Δεν ξέρω αυτή η έρευνα που θα μας οδηγούσε. Ως προς ε, θέματα ελέγχου συμφωνούμε ότι εδώ θα μπορούσαμε να ορίσουμε μία υποεπιτροπή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Επίσης, δεν θα πρέπει να επικρίνουμε τις ΙΠΑ σε ένα τέτοιο έγγραφο, τουλάχιστον όχι ε, με βάση πληροφορίες που προέρχονται από τον τύπο. Δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ πώς κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό. Πώς θα τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια. Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν θα δέχονταν κάτι τέτοιο, τουλάχιστον όχι πέραν ε, ενός ορίου. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να επιληθεί μέσω τροπολογιών, διότι θα πρέπει να έχουμε σαφείς απαντήσεις. Ο κύριος Γιάννιεθ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας με έχει ορίσει υπεύθυνο επί της έκθεσης αυτής. Κάθε φορά που μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εμείς δυστυχώς έχουμε μεγάλη πείρα. Υπάρχουν ε, βεβαίως και στοιχεία διαχωρισμού της τρομοκρατίας. Δεν πρέπει να τα συγχαίουμε. Νομίζω ότι η τρομοκρατία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας και για την ε, δημοκρατική μας κοινότητα. Γι' αυτό θα πρέπει σε κάθε έκθεση να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ συνέγραψα μία έκθεση στην προηγούμενη θητεία και σε κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Μιλάμε για τα αίτια της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν έχει αίτια, διότι αίτια σημαίνει ε, δικαιολογία. Δεν μπορούμε δηλαδή παρά να υποσκάψουμε αυτή την τάση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αίτια της τρομοκρατίας. Έτσι απλά υπάρχουν λέξεις παγίδες που θα πρέπει να αποφύγουμε. Δεύτερον, πρόκειται για μία μελέτη ή έρευνα σε σχέση με την τελευταία δεκαετία, μετά από το 9-11. Θα πρέπει την τελευταία πενταετία από το 2004-2005 μετά από τις τρομοκρατικές ενέργειες του Λονδίνου και της Μαδρίτης έχει μειωθεί ο αριθμός θυμάτων δραστικά. Αυτή η έκθεση αναφέρεται στην ορολογία της ε, Βορείου Αμερικής, δηλαδή της κυβέρνησης της Αμερικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας η παρούσα κυβέρνηση δεν το ορίζει με τα ίδια λόγια. γιατί όταν μιλάμε πόλεμος κατά της ε, τρομοκρατίας σημαίνει ότι δεχόμαστε τους πολεμοχαρείς ε, εκείνους τρομοκράτες σαν αντίπαλο δέος, κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει. Άρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί οι τρομοκρατικές ενέργειες και έχουν μειωθεί, έχει μειωθεί και ο αριθμός θυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουμε καταφέρει, ιδιαίτερα σε επίπεδο κρατών μελών. Και εδώ μιλώ για τον άκρατο Ισλαμικό, για την άκρατη Ισλαμική τρομοκρατία. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη άλλους πολιτισμούς, ιδιαίτερα το Ισλάμ. Γιατί δυστυχώς το ότι και ένα κοράνι στο Μαϊάμι οδήγησε στη δολοφονία υπαλλήλων των ΗΠΑ στο Πακιστάν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε όλες τις πτυχές της τρομοκρατίας, όλες τις διακλαδώσεις της. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μας ε, τρομάζει η λέξη καταστολή, γιατί όταν μιλάμε για τήρηση θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια κατασταλτική πολιτική για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας. Επίσης, ε, αυτό αφορά και την ε, χρηματοδότηση, κατάρτιση και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη δική μας πολιτική πολέμησης της τρομοκρατίας. Έχουμε μια παράδοση, ε, συγκεκριμένες αρχές, ένα αξιοκρατικό σύστημα και δεν μπορούμε να συγχαίουμε τη δική μας πολιτική με την αμερικανική πολιτική. Γιατί εμείς το Γκουαντάναμο το αντιμετωπίσαμε διαφορετικά. Υπάρχει ένα νομικό κενό, μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, Γκουαντάναμο. Αν και ορισμένες χώρες συνεργάστηκαν με την CIA κατά τις υπερπτήσεις καθώς και τα βασανιστήρια και τις ανακρίσεις. Υπήρχε δηλαδή συνέργεια. Αυτό σημαίνει ότι μέσω τροπολογιών μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο γιατί χρειάζεται μεγαλύτερη εμβάθυνση ιδιαίτερα ως προς το παρόν πλαίσιο της τρομοκρατίας. Ο κύριος ε, Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι πολύ ε, σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να πω στη Σοφή ότι δεν μπορώ παρά να τη συγχαρώ που αποτόλμησε να αντιμετωπίσει ένα θέμα τέτοιας εμβέλειας. Εγώ θεώρησα ότι υπήρχαν δύο οδοί αρχικά τον ε, δικό μας χάρτη όπως ισχύει ή να συνεισφέρω και εγώ με το μικρό μου ε, λιθαράκι. Ε, Σοφή, θα υποβάλω τροπολογίες, σου το λέω από τώρα να το ξέρεις, μερικές θα είναι προσθετικές και άλλες θα είναι τροπολογίες απαλυφής. Αλλά για να κρίνουμε την εμβέλεια της έκθεσης, για να την αποτιμήσουμε, θα πρέπει να ρωτήσουμε πόσα χρήματα δαπανούμε για την τρομοκρατία. Είναι αδύνατο να ποσοστοποιήσουμε κάτι τέτοιο και θα σας πω γιατί. Κάποτε στη χώρα μου, και αυτό είναι ένα παράδειγμα, ο που ε, κάθε εβδομάδα εδολοφονεί το ένας δημοτικός ε, σύμβουλος, είτε από πλευράς χριστιανοδημοκρατών, είτε από πλευράς σοσιαλιστών. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να προβάλλουμε ένα πλαίσιο προστασίας. Γιατί οι πολίτες που γνωρίζουν, που ζουν υπό συνεχή, συνεχές καθεστώς απειλής, πρέπει να προστατεύονται. Και αυτό αφορούσε και δημόσια προστασία αλλά και ιδιωτική. Πώς μπορούμε να ποσοστοποιήσουμε αυτή την προστασία, προστασία προσώπων, προστασία κτηρίων και ούτω καθεξής. Πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε την ωραία απασχόληση αυτών των προσώπων προστασίας, πόσες, ε, πώς, ε, πώς ορίζουμε την κοινωνική τους ασφάλιση. Πώς ορίζουμε την ε, προστασία με βάση ένα σύστημα πληροφοριών. Πώς ε, να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους, τους επιχειρηματίες, καθώς και τις ενώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις οικογένειες των θυμάτων. Πώς να αποτιμήσουμε τα χρήματα αυτά, τα οποία δίνουμε σε διπλούς πράκτορες. πώς μπορούμε να ορίσουμε τα χρήματα που δίνονται για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας ή ε, σε σχέση με εγκληματικές ενέργειες, την, ε, τα ναρκωτικά, τα οπλοστάσια που υπάρχουν, που προσπαθούμε να παροπλήσουμε, είναι αδύνατο να τα ποσοστοποιήσουμε όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, για ποια τρομοκρατία μιλάμε. Ο Λουίς είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Οι Ισλαμιστές ε, τρομοκράτες λένε ότι πρέπει να προσεύχονται να ε, ζητούν ανεξαρτησία και να κρατούν ένα όπλο στο χέρι. Πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα, γι' αυτό εύχομαι κάθε επιτυχία στη Σοφία με τα μικρά μου μέσα θα προσπαθήσω να τη βοηθήσω. Εγώ θα προβάλλω και ορισμένες προστίκες με τροπολογίες. Αλλά θα ήθελα να πω, Σοφή, ότι αναφέρθηκες και στην 11η Σεπτεμβρίου, αλλά θα πρέπει να αναφερθούμε στα θύματα, Σοφή, που είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα στα πλαίσια λήψης αποφάσεων, καθώς και στις τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν στην Ευρώπη, διότι θα πρέπει να προλαμβάνουμε και να προστατεύουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα συνεργαστώ μαζί σου με μια σειρά τροπολογιών που ελπίζω να λάβει σοβαρά υπόψη. Ευχαριστούμε κύριε Τίας Ντεμέρα. Επειδή μιλάμε για ευαίσθητα ζητήματα, θα πρέπει να είμαστε διεξοδικοί. Παρακαλώ λοιπόν, επειδή υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να μιλήσουν, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν χρονικά περιθώρια για να μπορέσουμε να έχουμε και τους τρεις προσκεκλημένους ομιλητές. Η κυρία Σίπελ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια όχι μόνο για το σχέδιο έκθεσης αλλά και για το πώς συζητήθηκε το θέμα. Σε πολλές συζητήσεις είχαμε την εντύπωση ότι μπορεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να κοστίζει οτιδήποτε χωρίς να έχει κανείς αντίρρηση και χωρίς να ζητάμε κάποιους υπολόγους. Το θέμα είναι ε, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το τι κοστίζει η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, μπορούμε, ε, όπως είπαν προηγούμενοι ομιλητές, ε, να έχουμε ε, κάποια όριστη εικόνα, αλλά έχουμε και πολύ συγκεκριμένα μέσα, γιατί έχουμε το SWIFT λόγω της τη Τρομοκρατία. Μιλάμε για το σύστημα στοιχείων επιβατών, το PNR, και πάλι λόγω της καταπολέμησης τρομοκρατία. Για να μην συζητήσουμε και τις δυνατό... Ε, τα στοιχεία που έχουν σχέση με την Europol κλπ. Έχουμε επίση ε, τα θέματα ελέγχου των υγρών στι πτήσει. Ε, όλα αυτά τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία αφορούν την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Πάρα πολλά μέσα, πάρα πολλέ πτυχέ που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό και για την συλλογή δεδομένων. Επίσης ε, είναι ευαίσθητο το θέμα και είπε πολύ σωστά ο κ. Σάλβαρο προηγουμένω ότι ε, θα πρέπει οι πολίτες να αποφασίζουν αν ε, θέλουν να δώσουν δεδομένα στο διαδίκτυο. Όμως ο κάθε πολίτης δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί με τα στοιχεία του. Δίνει τα στοιχεία του στην τράπεζα και δεν ξέρει για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν πολύ συχνά χρησιμοποιούνται επιπλέον δεδομένα ε, για σκοπούς για τους οποίους εγώ ως πολίτης δεν θα έδινα τη συγκαταθεσή μου. Όταν δίνω εγώ τα στοιχεία μου σε μια, εταιρεία, σε μια αεροπορική εταιρεία για να κάνει κράτηση της ε, θέσης μου σε μια πτήση, δεν δίνω στην εταιρεία τα στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσει για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα καθήκοντα τα οποία πρέπει να απαιτήσουμε και πρέπει συνεχώς να θέτουμε το ερώτημα για ποιους σκοπούς διατίθενται χρήματα και τι κονδύλια δίνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν συζητάμε πολύ συχνά τα αίτια της τρομοκρατίας και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα αίτια της τρομοκρατίας και τι μπορούμε να κάνουμε ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιοι θα είναι οι υποστηρικτέ μα για μια τέτοια συζήτηση. Ελπίζω, αν δεν το συζητάμε εμεί που είμαστε η Επιτροπή για τι εσωτερικέ υποθέσει, θα το συζητήσουν κάποιε άλλε επιτροπέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλέ ερωτήσει έχουν ήδη γίνει και έχουν δώσει ανάψματα για συζήτηση ε, που ε, θα χρειαζόμουν πολύ περισσότερο χρόνο. Θα προσπαθήσω να συντομεύσω όσο είναι δυνατόν, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να τηρήσω το όριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πρόταση, για το σχέδιο έκθεσης. Και εγώ ε, είμαι απόλυτα διατεθειμένος να συνεργαστώ για την καλύτερη διαμόρφωση του σχεδίου εκθέσεως. Εδώ δεν πρόκειται απλώς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή για θέματα ασφάλειας. Εδώ μιλάμε για αρχές του κράτους δικαίου, για κοινοβουλευτικό έλεγχο και κατά τη γνώμη μου στην τελευταία δεκαετία δεν δόθηκε επαρκή σημασία σε όλα αυτά τα θέματα ακριβώς λόγω της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ε, υπάρχουν θέματα λοιπόν ε, ε, κράτους δικαίου τα οποία ε, άπτονται της σφαίρας των ε, προσωπικών δεδομένων υπάρχουν και θέματα ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου τα οποία φύγονται λόγω της του αγώνα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας Πολύ συχνά υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στις συζητήσεις που γίνονται. Ξέρουμε ότι υπάρχουν θύματα από την τρομοκρατία και χρειάζεται καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Αλλά ε, θα πρέπει να λέμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι η τρομοκρατία ε, είναι ε, μια υποκατηγορία της εγκληματικότητας και τίποτα παραπάνω. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε με αποτελέσματα, να δούμε ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας μειώνονται και τα ποσοστά τρομοκρατίας όπως τα ποσοστά εγκληματικότητας. έχει βελτιωθεί η κατάσταση και νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να θέσουμε επιτάπητος και να τα συζητήσουμε αντικειμενικά. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται ε, να γίνει αυτό γιατί στα κοινοβούλια και στα εθνικά κοινοβούλια και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία δέκα χρόνια δεν τα συζητήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. όχι διότι πρόκειται για εθνικές αρμοδιότητες, γιατί πολύ συχνά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητάμε θέματα τρομοκρατίας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αυτό οδηγεί στο ότι έχουμε και αρμοδιότητα να ελέγχουμε τα μέτρα τα οποία θεσπίζουμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δύο σύντομες παρατηρήσεις τώρα που θεωρώ σημαντικές για την απόφαση πλαίσιο για την τρομοκρατία, για την οποία δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη έκθεση προς το παρόν, νομίζω ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα και για το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης. Χρειαζόμαστε σαφείς ορισμούς και πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τα θέματα τήρησης δεδομένων και με το θέμα της διαμόρφωσης εικόνας προσώπου, σκιαγράφησης προφίλ. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ορισμούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα με συγκεκριμένο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιμένω, είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα κάνουμε το καταδύναμη. Αλλά α είμαστε συνοπτικοί, λακωνικοί, για να βοηθήσουμε την ε, εισηγήτριά μα, την κυρία Ίνθβελτ να κάνει και δική τη δουλειά. Κύριε Ούλτβερτ, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε. Γι' αυτό θα είμαι όσο το δυνατό πιο σύντομο. Πρώτα απ' όλα εκτιμώ το έργο το οποίο έχει κάνει η Σοφή Ιντβελτ επειδή το θέμα παραμένει πολύ σημαντικό παρά το γεγονός που, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου φαίνεται ότι τα πράγματα είναι κάπως πιο ήρεμα. Αυτό είναι παραπλανητικό. Νομίζω ότι ε, πάντοτε θα υπάρξει έμπνευση για τους τρομοκράτες. Υπάρχουν αποθέματα εμπνεύσεων για αυτούς και θα αντιμετωπίσουμε φοβάμαι νέες προκλήσεις. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης και προσωπικά θα ήθελα να κάνω όχι 5 ως 10 παρατηρήσει, αλλά 3 ως 5 παρατηρήσεις, ή μάλλον τροπολογίες ε, σε ορισμένε παραγράφους εδώ. μαλλον τροπολογιες σε ορισμενε παραγράφου εδω η παραγραφος 7 στη σελίδα 6, κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντική, διότι καλεί την Επιτροπή να κάνει ένα χάρτη όλων των σημείων τρομοκρατίας στην Ευρώπη και ζητεί στα κράτη-μέλη να κάνουν αξιολόγηση όσον αφορά την αντιτρομοκρατικές τους πολιτικές. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα πολλά έγγραφα δεν δίνουν αρκετά στοιχεία σχετικά με τη ρίζα της τρομοκρατίας, για τη φύση της τρομοκρατίας, για τις διάφορες πηγές έμπνευσης της τρομοκρατίας, όπως και η τήσια έκθεση της Europol. Επειδή έχει πολλές στατιστικές, είναι φορτωμένη η έκθεση με πολλές στατιστικές και δυστυχώς δεν έχει ε, προγνώσεις, δεν έχει προβλέψεις σχετικά με τα γεγονότα που θα συμβούν, που μερικές φορές θα μπορούσαν να εκτιμηθούν εκ των προτέρων. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς όταν προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσα χρήματα ξοδεύουμε για την αντιτρομοκρατία. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να αναζητήσουμε και να βρούμε την απάντηση διαφορετικού ερωτήματος σχετικά με τι είδους γνώσεις συγκεντρώνομαι, τι αντιλήψεις υπάρχουν ε, μεταξύ μας, διότι είναι φανερό από τη συζήτηση που έγινε εδώ ότι συνήθως υπάρχουν οι δικές μας πηγές. Πρώτα απ' όλα τα έγγραφα, τα βιβλία, που είναι θεωρητικές αφηρημένες γνώσεις και δεύτερον η πραγματικότητα στις χώρες μας. Αυτή η έκθεση καλεί όλους μας να συνδυάσουμε αυτές τις δύο μορφές γνώσεων για να ενοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουμε για την τρομοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Στο τούρνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σοφή για την έκθεση αυτή και για την ακριβολογία που την διέπει. Ακούγοντας τα λόγια του κυρίου Γιάννη, συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο πως αυτά τα χρόνια, την τελευταία δεκαετία, στην Ευρώπη μιλάμε όχι μόνο για οργανωμένο έγκλημα, αλλά και ενισχυμένη τρομοκρατία που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Και αυτό το είδα και στη δική μου έκθεση και μέσα σε 10 χρόνια δεν βλέπω ποια ήταν τα απτά αποτελέσματα και τι ποσά δαπανήθηκαν. Κάτι το οποίο με εκπλήσει είναι ότι όλες μας οι ευρωπαϊκές πολιτικές καταπολέμησης τρομοκρατίας έγιναν διότι ε, αυτή ήταν η επιταγή των ΙΠΑ. Ε, είτε το αφορούσε το SWIFT είτε το TN, R, δηλαδή τα στοιχεία των επιβατών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μία διάκριση εδώ. Όταν μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορούμε να μιλάμε για την τρομοκρατία που αφορά τον ε, Ισλαμικό φονταμενταλισμό. Όμως υπάρχουν ε, διάφορες πηγές και τρόποι έκφρασης της τρομοκρατίας στη χώρα μου, στην Ιταλία. Η τρομοκρατία σκότωσε συνδικαλιστές, δημοσιογράφους, δίκαστες και μόνο το 2001 οι ερυθρές ταξιαρχίες μπήκαν στο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και λίγα χρόνια πριν ξανάρχισαν τη δραστηριότητά τους. Θα ήθελα λοιπόν να γίνουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν. Λοιπόν, η Προεδρία του Συμβουλίου είναι έτοιμη να κάνει μια παρατήρηση. Σας παρακαλώ να είσαστε πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε χρειάστηκε λίγος χρόνος για να συλλέξω τις ε, πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες για την εισηγήτρια πάλι το θέμα δεν είναι η αντιτρομοκρατία το βασικό μου θέμα. Γι' αυτό οι πληροφορίες μου δόθηκαν από συναδέλφους. Αλλά ίσως θα ήταν λογικό να σας δώσω μία σύνοψη σχετικά με το τι κάνει η Προεδρία σε αυτόν τον τομέα. Πρώτα απ' όλα υιοθετήσαμε συμμεράσμα του Συμβουλίου για την εσωτερική στρατηγική το Φεβρουάριο που καλύπτει και την αντιτρομοκρατία και προσπαθεί να καθορίσει το ρόλο των διαφόρων παραγόντων σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό, αν θέλετε, είναι ένα γενικό πλαίσιο που το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα ήθελαν να δουν μαζί στον, τομέα, στον ευρύτερο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Δεύτερον, η δική μας πρωτοβουλία για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της ασφάλειας. Ε, αναφερθήκατε σε αυτήν την άσκηση και ένα από τα απτά αποτελέσματα που ελπίζουμε να πετύχουμε είναι η οργάνωση της πρώτης συνάντησης πιέση και κόζη την 1η Ιουνίου και η αντιτρομοκρατία θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Ίσως, εάν σας ενδιαφέρει, θα μπορούσαμε να σας, δώσουμε, να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία της συνάντησης. Το τρίτο θέμα είναι οι δικαστικές πτυχές της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θα είδατε την έκθεση που είχε προετοιμαστεί από τον συντονιστή της αντιτρομοκρατίας και συζητήθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή του άρθρου 36. Και με αυτή τη βάση ε, τις επόμενες ημέρες θα το συζητήσει η Κόζη για να δει τις δικαστικές πτυχές που πρέπει να συζητηθούν από τις διοκτικές αρχές στην Ευρώπη και όπως είπα αυτό θα πάει στην, Κόζη μετά τις επόμενες δύο εβδομάδες και οι αντιπρόσωποι πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν με βάση αυτή την έκθεση που ετοίμασε ο συντονιστής αντιτρομοκρατίας. Ακόμα δύο παρατηρήσεις, θα είμαι σύντομος όμως. Ε, σκοπεύουμε να ετοιμάσουμε συμπεράσματα για τα βιολογικά πυρηνικά όπλα για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από διάφορες διακριτικές αρχές. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη σύνταξη των ε, συμπερασμάτων του Συμβουλίου, αλλά ε, ετοιμάζουμε συμπεράσματα στο Συμβούλιο. Και τέλος, η ασφάλεια της αεροπορίας, η Προεδρία τροφοδοτεί την αναθεώρηση των έξι μηνών που ετοιμάζει η Κομισιόν, η Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι η COSI είναι η στρατηγική κοινότητα η Στρατηγική Επιτροπή με συγχωρείτε στο Συμβούλιο που εξετάζει όλα αυτά τα ευρύτερα θέματα εσωτερική ασφάλεια και έχει εξοδοτηθεί να ενημερώνει από καιρού καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα όσα συζητούνται στην Επιτροπή. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη νομική υποχρέωση, με τα χαρά να σα στείλουμε και άλλε πληροφορίε για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τι διάφορε πρωτοβουλίε τι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Είχαμε αρκετές ε, παρεμβάσεις σημαντικές εδώ και τώρα η κυρία Ιντιβέλτ θα πρέπει να απαντήσει όχι στον καθένα αλλά παρακαλούμε να κάνει ορισμένε καταληκτικές παρατηρήσεις προτού ορίσουμε τις προθεσμίες για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν συντομότερη και να απαντήσω σε γενικές γραμμές στα βασικά θέματα που έθιξαν οι παρευρισκόμενοι. Ορισμένοι είπαν ότι δεν είναι εφικτό να γίνει ε, μια τέτοια άσκηση και να έχουμε την πλήρη εικόνα. Ίσως είναι σωστό αυτό που λέτε λόγω της φύσης ε, του θέματος και δεύτερον επειδή ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών αντιτρομοκρατίας ε, γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μα δεν είναι το θέμα του εφικτού, αλλά το θέμα τη ανάγκη, τη αναγκαιότητα. Το βασικό αντικείμενο τη αντιτρομοκρατική πολιτική είναι να προστατεύσει τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι προ το καλό της ε, δημοκρατία, του κράτου δικαίου και ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αξιολογούμε τα όσα έχουμε κάνει την τελευταία δεκαετία. Μιλάω για δεκαετία, αλλά ορθά μια συνάδελφος είπε ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρώπη ασχολούνται με αντιτρομοκρατικέ πολιτικέ εδώ και περισσότερο χρονικό διάστημα. Νομίζω όμω ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση μόλι ξεκινήσαμε να έχουμε κοινή ε, αντιτρομοκρατική πολιτική εδώ και μία δεκαετία. Επίση, απαντώ σε εκείνου που λένε ότι δεν πρέπει να επικρίνουμε τι ΗΠΑ στην έκθεση. Ναι και όχι. Το αντικείμενο της έκθεσης δεν είναι να επικρίνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το βασικό κίνητρο για τις αντιτρομοκρατικές μας πολιτικές τα τελευταία δέκα χρόνια προήλθαν από την 11η Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν απλά επίθεση στους Αμερικανούς, αλλά επίθεση στον τρόπο ζωής μας και ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούμε τον όρο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, υποστηρίξαμε τη στρατηγική τους ε, τα δέκα τελευταία χρόνια χωρίς να κάνουμε και πολλές ερωτήσεις. Υπό αυτή την έννοια, ακόμα και αν δεν είναι η πολιτική η δική μας, την αποδεχτήκαμε, την στηρίξαμε. Πάλι, το αντικείμενο της άσκησης. Ίσως δεν μπορούμε σε αυτή την πρώτη αξιολόγηση να τα δούμε όλα επιτάπητος και να έχουμε την πλήρη εικόνα. Αλλά νομίζω ότι καθήκον μας είναι ως κοινοβουλευτικό όργανο να έχουμε πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Και ο λόγος για τον οποίο έφτιαξα αυτή την έκθεση με αυτόν τον τρόπο είναι ότι είπα ξεκινήσουμε με ορισμένα συγκεκριμένα απλά ερωτήματα. Διότι αν πείτε για παράδειγμα, ότι χρειαζόμαστε κοινοβουλευτικό έλεγχο, πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Όλοι συμφωνούν σε γενικέ γραμμέ. Αλλά πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και να ζητούμε συγκεκριμένε απαντήσει. Ε, και Λότφορντ είπε ότι ε, πήραμε μια απόφαση. Και πού κατέληξε αυτό το μέτρο. Ε, αυτό είναι δύσκολο να θυμηθεί ποσοτικά. Πρώτα απ' όλα, γιατί τα κράτη-μέλη δεν απαντούν. Και δεύτερον, η Επιτροπή θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια άσκηση. Διότι αγαπητοί φίλοι, θέλω να πω το εξή. Το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, ζητώ συγγνώμη στον ε, καημένο εκπρόσωπο της Επιτροπής που αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει τη δουλειά της από την αρχή, τότε το Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνει πολύ ακριβούς συμβούλους για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ελπίζω στο μέλλον η Επιτροπή μόνη τη θα μα προσκομίσει αυτά τα στοιχεία. Τώρα, στο Συμβούλιο, σας είμαι ευγνώμων για τις παρατηρήσεις σας, αλλά νομίζω ότι μάλλον κοιτούσατε το μέλλον και τις νέες πρωτοβουλίες του Συμβουλίου, ενώ εμείς αυτό που κάνουμε είναι ε, βλέπουμε το παρελθόν. Βλέπουμε τι κάναμε τα τελευταία δέκα χρόνια και τι, ποια ήταν τα επιτεύγματα. Τι, πώς πρέπει να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας παρά ε, να βλέπουμε ότι υπάρχουν συνέχεια νέες πρωτοβουλίες ε, και να μην ξέρουμε πόσο αποτελεσματικές θα είναι. Μία από τις τελευταίες παρατηρήσεις ότι δεν υπάρχει αναφορά σε άλλες επιθέσεις παρά στην 11η Σεπτεμβρίου και στα θύματα. Όχι επειδή ε, τις έχω παραβλέψει αναφέρθηκα στις εθνικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο λόγος τον οποίο ξεχώρισα την 11η Σεπτεμβρίου είναι λόγω των επιπτώσεων που είχε για τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών αντιτρομοκρατίας. Επειδή αν θέλετε η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Ε, υπήρξε αντιτρομοκρατία εδώ και δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Βόρειο Ιρλανδία, Ελλάδα υπήρξε αντιτρομοκρατία. Δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά η 11η Σεπτεμβρίου ειλικρινά ε, επέφερε μια σημαντική αλλαγή. Νομίζω λοιπόν ότι έκανα τις παρατηρήσεις που έπρεπε να κάνω και προσβλέπω στις τροπολογίες σας και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα πριν από τις θερινές διακοπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ινβέλτ και όλοι καλείστε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας μέχρι τις 26 Απριλίου 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, γιατί έχουμε τρεις προσκεκλημένους ομιλητές που περιμένουν να λάβουν το λόγο. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν. Είναι ο κύριος Χίμπε από την Επιτροπή, ο κύριος Ράιτ που εκπροσωπεί την Europol και ο κύριος Breitbart Καλώ ήρθατε. Yes, I mean, it is important. It is important that we proceed. Πρέπει αμέσως να ξεκινήσουμε, χωρίς να καθυστερούμε γιατί ούτε μια ώρα δεν μας έχει μείνει. Μέχρι τις 6 και 30 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίασή μας. Μπορούμε βέβαια να ζητήσουμε ε, από τους διερμηνείς ε, να δείξουν γενναιοδορία. Θα κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε για να χρησιμοποιήσουμε τη μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μάλιστα για ένα ε, τόσο επίμαχο θέμα όπως είναι η εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Είναι το αποκαλούμενο πρόγραμμα TFTP και θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Rob Wainwright, διευθυντή της Europol τον κύριο Ράινχαρτ Πρίμπε που εκπροσωπεί το Διευθυντή Εσωτερικής Ασφάλειας της Επιτροπής και τον κύριο Πολ Μπράιτμπαρτ που εκπροσωπεί τον Ολλανδικό Φορέα Προστασίας Δεδομένων. Σας καλωσορίζω λοιπόν και τους τρεις. Και προτείνω να δώσουμε καταρχήν το λόγο στον κύριο Πρίμπε, μετά στον κύριο Βέινράιτ και τέλος στον κύριο Breitbart. και στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για τη συζήτηση. Σας παρακαλώ όμως για άλλη μια φορά να περιοριστείτε στο να κάνετε ερωτήσεις και να είστε σύντομοι. Κύριε Πρίμπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Η Επίτροπος Μάλστρομ παρουσίασε την αναθεώρηση ε, ε, ε, και την έκθεση της Επιτροπής το Μάρτιο και είπε η Επίτροπο ότι θα είναι διαθέσιμη για περαιτέρω διευκρινήσει αν χρειαστεί. Και εγώ ήρθα σήμερα εδώ για τυχόν διευκρινήσει που μπορεί να θέλετε. Αλλά και μετά τη σημερινή μα συνεδρίαση θα είμαι στη διάθεσή σα αν χρειαστείτε κάποιε διευκρινήσει. Μέσα σε έξι μήνε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτού του μηχανισμού. Οι μηχανισμοί βάσει τη συμφωνία έχουν υλοποιηθεί και η Επιτροπή έκανε κάποιες συστάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής της συμφωνίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 4, επαλήθευση, μηχανισμός επαλήθευσης, και είπε ξεκάθαρα η Επίτροπος ότι παρότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης εκτιμούμε την δουλειά που έχει γίνει από την Europol όσον αφορά την ε, υλοποίηση του τμήματο τη συμφωνία για το οποίο είναι υπεύθυνη. Ε, χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και να δώσουμε διευκρινήσει σε σχέση με το τι κάνει η Europol. Έχουμε δει ένα έγγραφο και θα το παρουσιάσει ο κύριος Wright και χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες το μηχανισμό επαλήθευσης. κατανοητό ότι μπορεί να υπάρχει πεδίο βελτιώσεων. Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα της πρώτης επιθεώρησης και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να, να το δούμε μετά από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να καταλήξουμε στο ότι η Europol έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά της ε, με επαρκή τρόπο. Με την GSP έχουμε συνεργαστεί επί 12 χρόνια για να εξασφαλίσουμε ένα πεδίο προστασίας δεδομένων και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ιδίως σε πολύπλοκα θέματα ούτως ώστε να καταλήξουμε σε κάποια κοινή θέση. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία τώρα βρισκόμαστε. Συνεργαζόμαστε, έχουμε ήδη κάνει ένα σεμινάριο και θα κάνουμε άλλο ένα το Μάιο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση για αυτό το θεμελιώδους σημασίας ε, θέμα όσον αφορά τη συμφωνία. Από το σημείωμά μας θα έχετε δει ότι δίνουμε υψηλή προτεραιότητα σε όλες τις συστάσεις του GSP και το βασικό θέμα μεταξύ Europol και GSP είναι η αρχή της αναλογικότητας ε, του άρθρου 4 και πώς πρέπει να λειτουργούν. ως θέμα προστασίας δεδομένων, ως επιχειρησιακό θέμα ή συνδυασμός των δύο είναι κυρίως ε, θέμα προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την GSP και δεν μας εκπλήσει αυτό γιατί η λειτουργία του GSP είναι ακριβώς το να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών ε, των θεμάτων ε, επεξεργασίας δεδομένων. Κατά τη γνώμη μου το άρθρο 4 προχωρεί και παραπέρα. Δεν είναι απλώς ένα συμβατικό άρθρο για την προστασία των δεδομένων. Η Europol είναι ιδιαίτερα πεπειραμένη στα θέματα προστασίας των δεδομένων. Έχουμε εμπειρία από τα περασμένα 12 χρόνια και ε, στη συμφωνία υπάρχουν όλα τα θέματα για την προστασία δεδομένων. Δεδομένα μόνο για περιορισμένο ε, με χαρακτήρα περιορισμένης επεξεργασίας. Υπάρχουν σαφείς διατάξεις για την διατήρηση και διαγραφή δεδομένων, για τη διαβίβαση δεδομένων για την ε, δυνατότητα πρόσβασης και για τη δυνατότητα ανάκλησης. Είναι πολύ ισχυρές οι διατάξεις ε, και τις εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας δουλειά. Σε ορισμένα θέματα ε, προχωρούν και παραπέρα από ότι είναι σύνθεση για τις συνήθεις αστυνομικές δραστηριότητες. Υπάρχουν ρήτρε σε άλλα σημεία της συμφωνίας και όχι στο άρθρο 4, συγκεκριμένα στο άρθρο 5, όπου υπάρχουν ειδικέ διατάξεις στις ΗΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις ειδικέ μνήες της ανταλλαγής δεδομένων Europol με τις ΗΠΑ, η, η λειτουργία της Europol με βάση τη συμφωνία δεν αφορά μόνο τις ρήτρες διασφάλισης προστασίας δεδομένων. Άρα με τα στοιχεία προστασίας δεδομένων άλλα 11 ε, άρθρα ε, εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο. Το άρθρο 4 αποτελεί μία ρήτρα διαφύλαξης έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα προσωρινά στοιχεία σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο προστασίας ε, δεδομένων. Άρα πρόκειται για ένα πιο περιορισμένο πουλ δεδομένων. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν συλλέγονται σε περιορισμένη αλλά παγκόσμια βάση. Γι' αυτό το άρθρο 4 μιλά για ε, ταύτιση δεδομένων έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, τρομοκρατία στο συνολικό της επίπεδο. Έτσι ορίζει η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Αυτό ορίστηκε και ε, σε σχέση με τη μεταφορά δεδομένων κατά την διαπραγμάτευση. Όμως η εφαρμογή του άρθρου 4 αυτής δεν σημαίνει ότι παραβιάζονται τα δεδομένα. Όποιος και να είναι ο όγκος των στοιχείων που μεταφέρονται δυνάμει του άρθρου 4 δεν μπορεί να γίνει από τις αρχές των ΙΠΑ τη στιγμή που υπάρχει η ρήτρα διαφύλαξης ή διασφάλισης για κάθε περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις δυνάμει του άρθρου 4 δεν είναι σημαντικές. Οι νομοθέτες θεώρησαν θα πρέπει να ισχύει ένα επιπρόσθετο μέτρο και όπως όρισε και η ομάδα αναθεώρησης, η Ενωμένη, η Ενωμένη Ευρώπη αναλαμβάνει πολύ σοβαρά αυτή την ευθύνη δυνάμει του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4 με βάση την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και μία εκτίμηση όχι μόνο υπό τη συμβατική έννοια του, του όρου της προστασίας δεδομένων, αλλά τι, του τι εννοεί είπα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε τις αποφάσεις, τις δικαστικές αποφάσεις για να ξέρουμε γιατί χρειάζονται επιπρόσθετες προσπάθειες ερμηνείας και καταπολέμησης, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την ανάλυση κινδύνου παρούσης και παρελθούσης τρομοκρατίας. Η Europol έχει αυτό το καθήκον γιατί χρησιμοποιούμε την πραγματογνωμοσύνη ανεξάρτητα δηλαδή χρησιμοποιούμε ε, εμπειρογνώμες που μπορούν να κρίνουν το θεμητό χαρακτήρα, την νομιμότητα των αιτημάτων των ΙΠΑ. Άρα ε, εξετάζουμε τις δικαστικές αποφάσεις κατά περίπτωση. Η συμφωνία ορίζει ένα πουλ δεδομένων που είναι αρκετά μεγάλο για να υποστηρίξει τον ερευνητή, αλλά στρίκτο σένσου και επιτρέπει την εξέταση σε αυτό το επίπεδο, διότι σε αυτό το επίπεδο ο ερευνητής δεν έχει προσβασιμότητα στα στοιχεία. Υπ' αυτή την έννοια ε, υπάρχει διαφορά αντιμετώπισης από το JSP και τη Europol γιατί θεωρούμε ότι το άρθρο 4 δεν αφορά ρήτρα διασφάλισης αλλά ε, ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο θα κρίνουμε οι ίδιοι. Άρα μιλάμε για ερμηνεία δυνάμει της νομικής υπηρεσίας κομισιών και ΕΠΑ, που είναι τα εμπλεκόμενα μέρη και όπως ορίζει και το Διοικητικό ε, Συμβούλιο της Europol. Δυστυχώς ε, τα αιτήματα των ΕΠΑ δεν είναι εμπεριστατωμένα όπως θα έπρεπε. Υπάρχει λάθος προσέγγιση ως προς τα oral reports. Έχουμε λάβει τρεις τέτοιους φακέλους εμπιστευτικού χαρακτήρα για καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας σε σχέση με, τα με το ίδιο το πρόγραμμα των ΗΠΑ η διαδικασία επαλήθευσης αφορά τα γραπτά στοιχεία που μας έχουν παρασχεθεί, τα οποία τεκμηριώνονται και συνήθως είπα, μας δίνουν ένα κείμενο 56 σελίδων, αριθμός που έχει αυξηθεί, επειδή ζητάμε πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία. Ποιες κατηγορίες καλύπτουμε, ποιο χρονικό διάστημα και, πιο, ποια γεωγραφική εμβέλεια. Άρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ε, γίνεται μία προσέγγιση στρίκτο σένσου. Στις πέντε υποθέσεις από τις οκτώ ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες πριν την επαλήθευση. Έχουμε διαδικασία επαλήθευσης της τεκμηρίωσης με βάση κάθε απόφαση που λαμβάνουμε και, και με βάση τα δεδομένα της νομικής υπηρεσίας. Έχουμε 80 σελίδες στο τέλος. Σύμφωνα με τις συμφωνίες μας μεταξύ ημών, κομισιών και ΕΠΑ, προσπαθούμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Χρειαστήκαν 16 μέρες σε μία περίπτωση, σε μία υπόθεση, γιατί υπήρχαν ε, περαιτέρω ερωτήσεις προς τη ΣΥΠΑ, ένα follow-up. Με βάση αυτά τα πλαίσια δεν, μπορεί, ε, δεν μπορούν οι ΥΠΑ να ισχυριστούν ότι είμαστε γραφειοκράτες. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να βελτιώσουμε τις εργασίες μας με την υποστήριξη της JSP και τις συστάσεις της. Μετά από την έκθεση θα γίνουν δύο σεμινάρια, έγινε ένα και θα γίνει άλλο ένα το Μάιο και ελπίζουμε να φτάσουμε σε μια καλύτερη κοινή θέση τους στις ε, επερχόμενες εβδομάδες. Ως προς το θέμα της διαφάνειας, σας είπα γιατί αυτή η τεκμηρίωση θεωρείται εμπιστευτικού χαρακτήρα από τη ΣΥΠΑ για να καλύψουμε και να προστατεύσουμε τον ευαίσθητο χαρακτήρα ετοιμάτων. Στη Europol έχουμε καθήκον να το τηρήσουμε αυτό και κατανοώ τις ανησυχίες των ΙΠΑ. Αυτό είναι ένα σημείο που αναγνωρίζουμε και στην έκθεση αναθεώρησης. Υπάρχει έλεγχος στη Europol, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπεθυριωτές της JSP δεν έχουν πρόσβαση παρά αυτές τις προαπαιτήσεις θεωρούμε ότι η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό θα έχουμε και έχουμε πάντα όλες τις πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν έχει αρθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας μεταξύ Europol και ΕΠΑ. Τέλος, Πρόεδρε, θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό καθήκον της Europol. Είναι στο ανώτατο σημείο της ιεράρχησής μας τους τελευταίους εννέου μήνες. Είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση και φαντάζομαι και η έκθεση αναθεώρησης το αναγνωρίζει αυτό, όπως είπε και η Επίτροπος Μάλμστρομ. Βεβαίως χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις και εργαζόμαστε για την εφαρμογή τους. Ελπίζω να κατανοείτε τις ε, δυσκολίες και τη δυσχέρεια του καθήκοντος, αλλά είμαστε ε, πλήρως δεσμευμένοι και θα σας απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Wainwright και πριν να ακούσουμε τις ερωτήσεις ε, των ευρωβουλευτών θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Breitbart που εκπροσωπεί τον Ολλανδικό Φορέα Προστασίας Δεδομένων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου δίνουν την ευκαιρία ε, να μιλήσω ενώπιόν σας. Εδώ εμφανίζομαι καταρχήν ως μέλος του κοινού εποπτικού φορέα, του JSB, στον οποίο συμμετέσχαν μαζί με τους άλλους εκπροσώπους προστασία δεδομένων ως εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ε, ταυτόχρονα έχω και το ρόλο ενός από τους συντάκτες της έκθεσης ε, τον Νοέμβριο. Ξεκινώ από την ε, κοινή ε, επιθεώρηση που έγινε. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από αυτό που έγινε. Οι Αμερικανοί παρουσίασαν μια ανοιχτή εικόνα αυτών που τους ενδιαφέρει, δηλαδή σε τι χρησιμεύει το πρόγραμμα και έχω πολύ λίγα να πω σε σχέση με την έκθεση αναθεώρησης. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της συμφωνίας που λεπτομερώς αναφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια μέτρα ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που προχωρούν περισσότερο από αυτά που γνωρίζουμε για την προστασία των δεδομένων. Συγκεκριμένα αυτό αφορά το ρόλο των ανεξάρτητων ελεγκτών που είναι πολύτιμο το έργο τους διότι παρακολουθούν προσεκτικά αυτό που κάνουν οι αναλυτές δεδομένων και προσπαθούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή να διακόψουν αυτή την ανάλυση αν κατά τη γνώμη τους δεν είναι βάσιμη η κατηγορία περί τρομοκρατίας. Είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Λιγότερο ευχαριστημένος είμαι με τον τρόπο με τον οποίο έχει συνταχθεί αυτή η έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκαν πολλές πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της δημοσίευσης αυτής της έκθεσης ε, στις αρχές Μαρτίου, αυτής της κοινή έκθεσης με την Europol. Ξεκινήσαμε αρχικά με το ότι η ομάδα των ε, ελεγκτών θα ασχολείται με την έκθεση αυτή πριν δημοσιευθεί, αλλά αυτό δεν έγινε. Στάλει μια πρώτη εκδοχή αυτής της έκθεσης σε όλα τα μέλη της ομάδας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά η έκθεση μετά τις τροποποιήσεις δεν διανεμήθηκε εκ νέου. Όντως θα μπορούσε να έχει κάποια ευαίσθητα στοιχεία. Πάντως, ε, επί αυτής της βάσης το στείλαμε στους Αμερικανούς συναδέλφους για να το εξετάσουν ε, και να, το, και να μπορούν ε, να αφαιρέσουν κάποια στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα. Μετά τις 8 Μαρτίου η Επιτροπή έστειλε συστημένη αυτή την έκθεση στα μέλη της Επιτροπής επιθεώρησης αλλά την έκθεση αυτή στις κάτω χώρες ε, εμείς την είδαμε αργότερα αφού πρώτα είχε παρουσιαστεί σε εσά την Επιτροπή και αφού επιμείναμε πολύ στις 15 Μαρτίου και μετά από έγκριση των Αμερικανών τότε στάλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυτή η έκθεση αλλά μόνο λίγες ώρες είχαν μείνει πια για να μπορέσουμε να δώσουμε τη θέση μας για αυτό το κείμενο. Μα είπαν ότι είναι πολύ ευαίσθητο πολιτικά το θέμα και δεν μπορούμε να δεχτούμε τις σα γιατί ήδη η Επίτροπος έχει δώσει το πράσινο φως και είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να τροποποιηθούν μέσα σε αυτήν την έκθεση. Συγκεκριμένα οι αποδείξει που πρέπει να δίδονται για τον σημαντικό χαρακτήρα των στοιχείων τύπου TFTP. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να εξηγήσουν τον χαρακτήρα αυτών των δεδομένων και μα ανέφεραν συγκεκριμένα παραδείγματα και καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό στην πράξη για του Αμερικανού. Όμω δεν έχω πιστεί για τη χρησιμότητα, για τη σημασία αυτών των δεδομένων. Δεύτερον, όσον αφορά τα δικαιώματα των εμπλεκομένων, ε, όντω τηρήσαμε τι απαιτήσει τη συνθήκη, αλλά όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, διότι τα εν λόγω άτομα δεν μπορούν να ζητήσουν διόρθωση αυτών των στοιχείων παρά μόνο για τα στοιχεία τα οποία ήδη αναλύθηκαν από τους εμπειρογνώμονες των Αμερικανών και αναφέρονται στην έκθεση της ε, κοινή ε, Επιτροπής ε, Επιθεώρησης πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να εκφράσω ως κριτική ε, είναι το συμπέρασμα που αναφέρεται για το ρόλο της Europol. Ίσως εκφράζεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Αυτή η έκθεση της, του JSB, του Κοινού Εποπτικού Φορέα, ε, εκφράζει κάποια κριτική για το ρόλο της Europol ε, και σε πολλές άλλες εκθέσεις βλέπω ότι η Europol αποφάσισε να διορθώσει κάποιες διαδικασίες. Διαπιστώνω ότι και οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ότι χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε γραπτώ για να μπορούμε να αιτιολογήσουμε κάποια αιτήματα. Όμω ο τρόπο με τον οποίο αυτό εμφανίζεται μέσα στην έκθεση επιθεώρηση δίνει μια χρειά ιδιαίτερα θετική. Δεν ξέρω σε τι βασίζεται αυτή η έκθεση, γιατί η ομάδα τη επιθεώρηση συζήτησε επί μία ώρα, είδε μόνο μία επιστολή τη Γυροπόλ για τη μέθοδο εργασία και μόνο για την αμερικανική μέθοδο ε, μιλούσε αυτό το ερώτημα. Ίσως να ξανασυζητήθηκε με την Europol, αλλά δεν συζητήθηκε με ολόκληρη την ομάδα των ε, εποπτών. Τώρα όσον αφορά την Europol, Υπάρχει μια λεπτομερή συζήτηση στην ομάδα εργασία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ράιτ και το θέμα είναι αν το άρθρο 4 περιλαμβάνει μια ρήτρα προστασίας και αν ε, είναι λειτουργική αυτή η ρήτρα. Πρέπει να μιλήσουμε για την προστασία των δεδομένων. Αυτό ήδη υπάρχει στην αιτιολογική σχέση και το άρθρο 1 αρχίζει να μιλά για τον ιδιωτικό χαρακτήρα και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Μιλάμε λοιπόν για τα προσωπικά δεδομένα και τραπεζικά δεδομένα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να συνεχιστεί με τη Europol και με τον κοινό υποπτικό φορέα JSP για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ. Τώρα, οι ερωτήσει. Κύριε Γουσοτήλ, παρακαλώ. Είναι θέμα διαδικασία. Ναι, είναι θέμα διαδικασία. Υπό το φω των δηλώσεων που έγιναν από τον τελευταίο μιλητή και οι σοβαρές ανησυχίες ε, που διατύπωσε, θα πρέπει να έχουμε ε, μία αντίδραση από την έδρα πρωτού παρέμβουμε, ότι αυτές οι ανησυχίες θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Ε, Είχα την πρόθεση να κρατήσω λίγο χρόνο για τις απαντήσεις. Πρώτα ακούμε τις ερωτήσεις, θα ακούσουμε τις ερωτήσεις αλλά να αφήσουμε λίγο χρόνο για αντίδραση από την έδρα, από τους ομιλητές. Λοιπόν, αν θέλετε να απαντήσουν πρώτα στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και μετά να γίνει δεύτερος γύρος ερωτήσεων. διότι Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Διαφορετικά ε, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Εκπλήσω με τα όσα άκουσα από τον κ. Blackbart. Θα ήθελα να είμαι απόλυτα σαφής η Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση για την αναθεώρηση και είμαι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μιλήσει για αυτή την έκθεση. Η έκθεση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή αφού είχε την έγκριση όλων των μελών της ομάδας. Και αν τώρα αμφισβητείτε, αυτό είναι ένα σημαντικό προηγούμενο, είναι ένα συμβάν σημαντικό. Αυτό όμως δεν ήταν αυτό που πιστεύαμε όταν η Επιτροπή έκανε, ε, ε, ε, την έκθεση. Και όλα τα μέλη της ομάδας αναθεώρησης συμφώνησαν και ο κύριος Βράιπαν ο ίδιος έκανε ορισμένες παρατηρήσεις για τη διατύπωση της έκθεσης. Και το 98% από ό,τι θυμάμαι είχαν ληφθεί υπόψη. Και θα μπορούσα όχι τώρα αλλά αργότερα να σας πω ε, σε ποια σημεία είχαμε συμφωνήσει. Λοιπόν, εκπλήσω με ειλικρινά, είναι κάτι το ε, ασύνηθες. Αλλά αν κάποιο μέλος από την ομάδα μπορεί ε, να μας μιλήσει ή κάποιο μέλος έχει αντίρρηση, τότε είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό μας. Τα άλλα μέλη της ομάδας αναθεώρησης, ακόμα και οι εκπρόσωποι της προστασίας των δεδομένων, συμφωνήσαν και εξακολουθούν να συμφωνούν με την έκθεση. Θα κάνουμε το γύρο των ερωτήσεων έτσι ώστε να έχουμε ένα λεπτό για τις απαντήσεις. Σας έλεγα ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο για τις απαντήσεις. Ο κύριος Άλβαρο. Θα ήθελα να ότι αν συμφωνούν οι συνάδελφοι μπορούμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Διότι βεβαίω ε, οι Γερμανοί θα πρέπει να αποχωρήσουν. Αυτό όμω δεν μα σταματάει από το να συνεχίσουμε εμεί. Λοιπόν, εάν ένα πράγμα είναι σαφέ, ανεξάρτητα με το τι υπόθηκε εδώ, ένα πράγμα είναι σαφέ. Ότι το πρόβλημα δεν είναι η Europol. Θα ήθελα να το πω αυτό, κύριε Γουαρμάιν, διότι το είπα και δημοσίω. Αν είναι πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε αν είσαστε το σωστό πρόσωπο, σωστή θέση. Είπατε, εγώ δεν έχω, είπατε ότι δεν έχετε πρόβλημα με τη Europol, διότι στη σελίδα 11 της έκθεσής σας δηλώνεται ότι η Europol ακολουθεί την ερμηνεία τη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σα λέει πώ θα ερμηνεύσετε το άρθρο 4 τις συμφωνίες και μπορεί εδώ να υπάρχει διαφορετική ερμηνεία μεταξύ μας διότι είναι δύσκολο να δούμε κατά πόσον αυτό είναι ένα λειτουργικό άρθρο ή αναφέρει την προστασία των δεδομένων αλλά το θέμα είναι ότι περιλαμβάνει και πλευρέ τη προστασία δεδομένων. Εάν η Επιτροπή δεν δέχεται ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο τη προστασία δεδομένων, ε, ε, ε, μιλούσαμε διαφορετική γλώσσα. Διότι το άρθρο 4.2 παρουσιάζει βασικά πράγματα. Αν θέλετε να έχετε προστασία δεδομένων. Το ζητούμενο είναι ότι ο προσδιορισμός είναι σαφές και η ανάγκη των δεδομένων ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι σαφή. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ε, ε, σκοπός να περιοριστεί η ροή δεδομένων προς τις Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να αποφύγουμε ε, την ε, μεταφορά των δεδομένων, αλλά κατέργωση των δεδομένων, αλλά αυτό δεν σημαίνει Γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια για να μην ε, ελαχιστοποιηθούν αυτά τα δεδομένα που στέλνονται στη ΣΥΠΑ. Τώρα, στην αναθεώρηση της συμφωνίας πρέπει να πούμε ότι υπήρξε περιορισμός των δεδομένων, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ποιο ποσοστό. Τώρα, τα διάφορα θέματα και ζητώ ε, συγγνώμη που δεν μπορώ σε 20 δευτερόλεπτα να απαντήσω. Το άρθρο 13 της συμφωνίας ορίζει ότι στην αναθεώρηση ε, υπήρξαν μηνύματα ε, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται. Αυτό όμως δεν προβλέπεται στη συμφωνία. Και επειδή η Europol δεν μπορεί να γνωρίζει, δεν σημαίνει ότι και η εταιρεία SWIFT δεν μπορεί να ξέρει. Και αν η εταιρεία, ε, ε με σχόλια, αν η Επιτροπή κάνει ε, μια έρευνα και αν θέλει να, να συνεργαστεί η SWIFT, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι αριθμοί. Εάν συνεργάζεται η SWIFT να το γνωρίζουμε. Τουλάχιστον στα δημόσια θέματα ε, νομίζω ότι θεωρείται ότι συνεργάζεται. Το ερώτημα είναι ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ άρθρου 4 και 5. Το άρθρο 4 ε, δεν αναφέρεται μόνο στη δημοκρατία, αλλά οι ορισμοί εξηγούν ότι είναι ανάγκη να υπάρξει σαφής προσδιορισμός και εξηγούν τις σχέσεις. Δηλαδή, θα ήθελα η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, να παροτρύνει ε, το Υπουργείο Οικονομικών να προωθήσει ε, στη Europol αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους δικούς μας οι στην Europol. Εάν θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ τους. Αλλά ε, στην έκθεση αναθεώρησης αναφέρονται πάνω από 20.000 αναζητήσεις. Δηλαδή 6-6 μήνες είχαμε 146 ε, αναζητήσεις την ημέρα. Δεν μπορώ πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε με, ένα τέτοιο, με μια τέτοια ποσότητα αναζητήσεων. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Αναφέρεται, αναφέρονται 304 αναζητήσεις, δηλαδή 1,2% όλων των αναζητήσεων. Λιγότερο και από στατιστικά στοιχεία. Εάν λοιπόν αυτό το βλέπουμε, ε, το έχουμε πάρει σοβαρά, θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Τώρα, για τις απαιτήσει προστασίας δεδομένων, κυρίως στα άρθρα 15 και 16, η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι η ε, Υπουργείο εξηγεί ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αρκετά οι δυνατότητες να ε, ασκηθούν τα, δικαιώματα προστασίας δεδομένων γνωρίζω γιατί δεν απήντησε το Υπουργείο. Θα έπρεπε να γνωρίζουμε όμως γιατί οι εθνικές υπηρεσίες προστασίας δεδομένων δεν έχουν απαντήσει. Και κάτι το πολύ ενδιαφέρον, επειδή αυτό παραβιάζει το άρθρο 16, αναφέρεται ότι οι μόνες αλλαγές που μπορούν να γίνουν στην βάση δεδομένων TFT είναι οι συνέπειες μιας ενημερωμένης, ενός ενημερωμένου αρχείου Δηλαδή οι τράπεζες είναι εκείνες, όπως αναφέρει η έκθεση, οι οποίες θα πρέπει να στείλουν μια διόρθωση των δεδομένων που ουσιαστικά που δεν συμφωνεί με το άρθρο 16. Αυτά είναι λίγα από τα θέματα όπου δεν υπάρχει συμβατότητα με τη συμφωνία. Δύο θέματα που αφορούν την Europol. Επειδή διαβάσαμε αυτή την έκθεση και ευχαριστούμε που καταβάλατε αυτή την προσπάθεια για να παρουσιάσετε συνοπτικά την έκθεση. Η συμφωνία λοιπόν ορίζει ότι ε, ένα αίτημα πρέπει να προσδιοριστεί το ταχύτερο δυνατόν για να γνωρίζουμε ποια είναι τα δεδομένα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και οι τεχνικές διαδικασίες απαιτούν να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι τρομοκρατίας. Η συμφωνία όμως έχει ως τίτλο ε, χρηματοδότηση και ε, αναζήτηση τρομοκρατίας. Πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος του τίματος, εφόσον μιλάμε για το πρόγραμμα ανείχνευσης τρομοκρατίας. Το άλλο, για το bulk, και αυτό είναι πολύ περιορισμένο το βρήκαμε στην έκθεση Europol, μαζική μεταφορά δεδομένων. Οι αρχές έδειξαν ότι στις ε, αναζητήσεις, στις ε, αναζητήσεις, είναι δυνατόν να γίνει και η μεταφορά αυτών των δεδομένων. Και θα, αυτό δεν σημαίνει ότι ζητούμε ε, τα δεδομένα από όλες τις χώρες καταλήγω λέγοντας ότι πιστεύω ότι η αναθεώρηση της συμφωνίας θα γίνει σε 1,5 χρόνο. Θα ήθελα να γνωρίζω από ένα τρίτο φορέα, από κάποιον ο οποίος είναι νομικά ανεξάρτητος, να μας πει κατά πόσον η υλοποίηση μέχρι τώρα συμφωνεί από νομικής απόψεως με την συμφωνία και πού βασίζονται αυτές οι εκθέσεις. Και πρέπει να σκεφτούμε να αναστείλουμε τη συμφωνία διότι προφανώς φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση στην εφαρμογή παρά σαφήνεια. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να αναφέρω. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι η τελευταία φορά που θα το συζητήσουμε. Απλά θα ήθελα να σας πω ότι ε, πραγματικά μας ανησυχεί αυτό. Μας ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται. Επειδή φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο εμπιστεύθηκε στη συνεργασία που είχαμε με τις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας για τους πολίτες μας στην εσωτερική ασφάλεια, ενισχύοντας όμως και το δικαίωμά τους ε, για να ελέγξουν κατά πόσον όλα γίνονται καλά. Και έχουμε την εντύπωση ότι αυτά δεν έχουν γίνει και δεν μπορείτε να περπατάτε με το ένα πόδι. Ωραία για τον εισηγητή. Έχουμε και το σκιώδη εισηγητή. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Όχι μόνο για τους διερμηνείς, γιατί όλοι έχουν άλλες υποχρεώσεις μετά τις 6.30 και οι προσκεκλημένοι μας ομιλητές. Όλοι έχουν κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις που πρέπει να σεβαστούμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις για να μπορούν να δοθούν και συγκεκριμένες απαντήσεις. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αλλά έχει τύχει και στο παρελθόν όταν υπάρχουν τόσο ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις ε, να τους δίνεται λίγο περισσότερος χρόνος. Ήδη ανέφερε ο κύριος Άλβαρο αρκετά. Θα ήθελα να κάνω μια βασική παρατήρηση. Μετά την συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούσε η διαδικασία του SWIFT να αποτελέσει ένα μήνυμα για αυξανόμενο σεβασμό και καλύτερη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς ε, δεν έγιναν καθόλου έτσι τα πράγματα. Υπάρχει δυσπιστία όσον αφορά τις, ε, τα ευρωπαϊκά όργανα και όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι λυπηρό όχι μόνο για αυτή τη συμφωνία, αλλά και για την εμπιστοσύνη την οποία μπορούν να έχουν και άλλες συμφωνίες και υπονομεύει ε, την ασφάλεια την οποία θα θέλαμε να έχουμε από τέτοιες συμφωνίες. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο και δραματικό σε σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Και στις διαπραγματεύσει, αλλά και στην συνθήκη και στη συμφωνία ζήτησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε με βάση τις κατηγορίες ε, του SWIFT να ακολουθήσουν μια πολύ στενή προσέγγιση Ακούσαμε από τον κύριο Γουέν Ράιτ ότι δεν τηρήθηκε. Χρειάστηκαν 16 μέρες για την απάντηση και χρειαζόντουσαν συνεχώς ε, να δίδονται νέες ερωτήσεις και απαντήσεις. Παραμένει το ερώτημα αν αυτές ε, οι προφορικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που μπορεί να είναι γραπτές ε, ή προφορικές. Παραμένει επίσης αβεβαιότητα για το ποια είναι η αρχική βάση. Η βάση είναι ε, ε, ε, κάποιο ύποπτο άτομο ή είναι ένα γενικό αίτημα. Μπορεί να υπάρχει ένα όριστο αίτημα για το οποίο δεν δίδονται συγκεκριμένα στοιχεία και η κυρία Μάλιστον είχε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αίτημα και ενδεχομένω ε, με συγκεκριμένο όνομα. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, να μπορούν ε, ε, να ακολουθούν συγκεκριμένου κανόνε για το τι μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω τη Συμφωνίας. Ποια είναι τα συγκεκριμένα αιτήματα που μπορούν να γίνονται και πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση των δεδομένων που τηρούνται. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για να έχουμε εμπιστοσύνη και σε επόμενες μελλοντικές συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η συμφωνία. Είναι κάτι στο οποίο συμφωνήσαμε και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί σωστά. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα. Σε δύο σημεία του κυρίου Wainwright θέλω περισσότερε διευκρινήσει, γιατί δεν τα θεώρησα απόλυτα πιστικά. Είπατε ότι το άρθρο 4 δεν είναι μια ρήτρα προστασία δεδομένων με εκπλήσει αυτή σας η θέση, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι. Και όταν συμφωνήσαμε, αυτό είχαμε κατά νου. Θα ήθελα λοιπόν μια λεπτομερέστερη εξήγηση αυτού που μας είπατε. Δεύτερον, για τις προφορικές πληροφορίες και ανταλλαγές πληροφοριών, και εδώ δεν είμαι πεπισμένος. Οι προφορικές ανταλλαγές πληροφοριών αποτελούν συμπληρωματικό αίτημα το οποίο απαντάτε προφορικά ή όχι δεν πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται με διαφορετικό τρόπο, με τρόπο που θα προστατεύει καλύτερα την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ, κύριε Διαθεμέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέχομαι τις ε, εξηγήσει και τις διευκρινήσεις του Διευθυντή της Europol για την εφαρμογή της συμφωνίας και γνωρίζω τις ε, δυσκολίες που γνώρισε για να φέρει σε πέρας το περιεχόμενο του άρθρου 4. Εκεί που δεν συμφωνώ είναι στη, ως προς την θέση της ε, κοινή εποπτικής αρχής. Η κοινή εποπτική αρχή δεν, ε, δεν εκπλήρωσε σωστά την εργασία της. Δηλαδή στο, στις 27 Μαρτίου άρχισε ένα διάλογο χωρίς να λάβει υπόψη τη Europol, την Κομισιόν και τις αρχές των ΙΠΑ. Ε, αντιβαίνοντας το άρθρο 13, διότι το άρθρο 13 μιλά για την κοινή αναθεώρηση με την κυβέρνηση των ΙΠΑ. Αυτό είναι πρωτοφανές το άρθρο 4 ζητά από τη Europol να επαληθεύσει ότι κάθε αίτημα αφορά περιοριστικά τα στοιχεία που ζητούνται, συσταλτικά δηλαδή. Άρα θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη το άρθρο 4, διότι το TFTP, η χνηλάτιση αυτή, δεν αφορά τα στοιχεία που προέρχονται από τον φορέα SWIFT ως προς την προστασία δεδομένων TFTP πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Μετά από ενδελεχή έρευνα. Άρα ο εκπρόσωπος της κοινή εποπτικής αρχής κάνει λάθος γιατί μιλά για στοιχεία του TFTP που ε, ελέγχει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ε, Δεδομένων. Μιλάμε για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό δεν είναι θέμα που αφορά αρμοδιότητα της κοινή εποπτικής αρχής. Και από την άλλη πλευρά, η Europol έχει λάβει 8 αιτήματα. Το τελευταίο το έλαβε στις 8 Μαρτίου. Από τα 8 αιτήματα ε, ζητήθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες ε, στα τέσσερα. Αυτό το σύστημα πρέπει να διευθετηθεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία δεδομένων με βάση αυτές τις εκθέσεις που είναι πολύ Και επίσης ένα μήνυμα προς την κοινή εποπτική αρχή. Η Europol, δυνάμει του άρθρου 4, ζήτησε την ισχύ εμπιστευτικού χαρακτήρα των εκθέσεων το Νοέμβριο του 2010 με βάση τις αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ζήτησαν οι αρμόδιες αρχές. Κύριε υπεύθυνε της κοινή εποπτικής αρχής, είχατε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, ακόμα και ε, σε εκείνα που φέρουν την μνήμα UE Secret. Η Europol έδωσε στοιχεία στα Κάτς και Κόζη και έδωσε πληροφορίες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις 31 Ιανουαρίου. Θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε όλες τις μεθόδους και τις διαδικασίες. Αλλά δεν συμφωνώ ούτε συμμερίζομαι την ιδέα ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα συστήματα της κοινή εποπτικής αρχής έξι μήνες μετά από την συμφωνία. Η κυρία Αντιβενότ. Okay. Then, Mrs. Albrecht. Κύριε Albrecht, παρακαλώ. Ο κύριος Albrecht. Ένα λεπτό μόνο. Νομίζω ότι αυτά τώρα τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε ενώπιόν μας δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με τότε που επαναδιαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία. Είχαμε τότε λίγες περιπτώσεις μεταβίβασης δεδομένων με πολύ στενή αντιμετώπιση, ελεγχόμενα με έναν ανεξάρτητο επόπτη. Τώρα έχουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών που εστάλησαν στις ΗΠΑ χωρίς δυνατότητα στενής αντιμετώπισης και έχουμε έναν επόπτη που έχει δει μόνο μικρό ποσοστό περιπτώσεων αναζήτησης και δεν έχει τη λειτουργία ενός ε, ανεξάρτητου επόπτη. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου αυτό που είχαμε κατά νου ότι θα συνέβαινε και πιστεύω ότι δεν άλλαξε τίποτα από τη στιγμή πριν από τη συμφωνία. Και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι για μένα που ε, υπερασπίζομαι το κράτος δικαίου ε, ε, εάν δεν μπορείς να αποδείξεις ότι μπορείς να ελέγξεις αυτές τις διασφαλίσεις και να επιβάλλεις αυτά τα μέτρα τότε θα πρέπει να σταματήσουν οι, αυτές ε, οι παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Wainwright και μετά στον κύριο Πρίμπε και μετά στον κύριο Breitbart. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω συντομία σε τρία σημεία. Πρώτον, όσον αφορά το δίκτυο τρομοκρατίας ε, και αυτό που ανέφερε ο κύριος Άλβαρο για το νέξους ε, τρομοκρατίας, θα πρέπει ε, να υπάρχει ένα τέτοιο νέξους και ιδίως όσον αφορά το COFOR. Υπάρχουν συγκεκριμένες έρευνες για συγκεκριμένα ονόματα και ε, αυτό δεν είναι θέμα του άρθρου 4 και μόνο. Νομίζω ότι ακολούθησε πολύ αργότερα στη συμφωνία. Αλλά ιδίω με βάση το άρθρο 4 ε, για τη μεταβίβαση, για τη μαθητική μεταφορά δεδομένων, θα πρέπει να ισχύσει και οι ΗΠΑ θα πρέπει να πείσουν την Europol γιατί υπάρχει στον κατάλογο η Α και όχι η Β χώρα. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε το ιστορικό, γιατί η Α χώρα είναι πιο συγκεκριμένη, στο, πιο σημαντική στο δίκτυο τρομοκρατίας, ίσως γιατί έχει ένα ιστορικό τρομοκρατίας ή κάτι άλλο. Ε, αυτό είναι σαν απάντηση του, ε, γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις επιμένουμε και σε άλλε όχι. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία προσπαθούμε να εντοπίσουμε υπόπτους τρομοκρατίας. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν συνεχίζουμε να έχουμε υπηρεσίε του Nexus. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μια στενή αντιμετώπιση. Δεν συμφωνώ με σας κύριε Άλμπρεχτ. Η διατύπωση για την ε, στενή αντιμετώπιση, για την αντιμετώπιση υπό τη στενή έννοια, είναι μια διατύπωση που επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Κατά τη γνώμη μου είμαστε ικανοποιημένοι ότι όντως έχουμε ακολουθήσει την αντιμετώπιση υπό τη στενή έννοια. Προς τον κύριο Μπουζουτήλ, που κάνατε δύο πολύ καλές ερωτήσει. Καταρχήν για την προστασία δεδομένων. Δεν υπάρχει ιδιαίτερα προστασία δεδομένων. Να σας πω τι εννοώ. Πολύ, με πολύ τεχνικά, τεχνικούς όρους εφαρμόζουμε αυτά τα μέτρα όταν εντοπίζονται κάποια συγκεκριμένα άτομα, αλλά δεν εντοπίζονται κάποια άτομα στο πλαίσιο του άρθρου 4. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακολουθεί. Τούτου λεχθέντος συμφωνώ με τον κύριο Άλβαρο ότι η όλη συμφωνία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει γενικές αρχές της προστασίας των δεδομένων. Και έμεσα και όσον αφορά το άρθρο 4 εφαρμόζουμε την αρχή της αναλογικότητας. Εδώ συμφωνώ απολύτω. Για τη δεύτερη ερώτησή σα τώρα για την προφορική ανταλλαγή δεδομένων. Έχουμε στενή σχέση συνεργασία με τους εταίρους μας στι ΗΠΑ και σχεδόν καθημερινά επικοινωνούμε και αυτό είναι ε, φυσιολογικό πέραν τούτου, σε πλαίσιο απόρριτων συνομιλιών, ε, έχουμε ε, συζητήσεις ε, για συγκεκριμένα στοιχεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο των ετοιμάτων του άρθρου 4, χρειάζονται επίσημες αποφάσεις επαλήθευση. και εκεί πάντοτε βασιζόμαστε στο έντυπο των 80 σελίδων που έχουμε. Νομίζω ότι δεν το εξηγήσαμε στην JSB, στην Κοινή Εποπτική Αρχή. Κακώ δεν το εξηγήσαμε, ήταν δικό μα φάλμα και έχει δίκιο η JSB που το αναφέρει στην έκθεσή τη. Τώρα όμω νομίζω ότι ε, είναι, έχει διευκρινιστεί η κατάσταση και ελπίζω στου επόμενου μήνε να είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτά ήταν τα τρία σημεία στα οποία ήθελα να αναφερθώ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρίμπε. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν τελειώνει ποτέ ο διάλογος όσον αφορά την ερμηνεία της συμφωνίας. Νομίζω ότι πολλά είναι σχετικά. Επαναλαμβάνω τα όσα είπε η Επιτροπή πριν από τα συμπεράσματα, μετά και αυτό, αυτή η συμφωνία αφορά τη μεταφορά των δεδομένων. Επίσης αναφέρθηκε σαφέστατα ότι θεωρούμε ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Αναγκάσαμε δηλαδή, τους Αμερικανούς να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει πρόοδος, συνεπώ παρά τι ε, αμφιβητήσει σα. Αλλά, επίση είπαμε, ότι αυτό περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και όχι μόνο εκείνα που ε, δόθηκαν στα πλαίσια της ε, συμφωνίας TFP, αλλά περιλαμβάνονται στοιχεία, δεδομένα και άλλων χωρών και το σημαντικότερο αμερικανικά δεδομένα. Επίσης, και αυτό συμβαίνει συχνά, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά εκτίματα για το ίδιο άτομο. Αυτό το οποίο μας είπαν οι Αμερικανικές αρχές είναι ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή έναν τρόπο να κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των αναζητήσεων ε, και να ξέρουν ποια, ε, ποιες γίνονται στα πλαίσια του TFTP. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες που δημιουργούν σύγχυση αντί να ε, διευκρινίζουν τα πράγματα. Στην τελευταία ε, φράση η έκθεση λέει θα γίνει μια αναθεώρηση του χρόνου. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Αντάβο πιστεύει θα γίνει σε 1,5 χρόνο. Θα γίνει μεταξύ 1ης Πρώτου και 31 Δωδεκάτου του χρόνου. Ευχαριστώ. Κύριο Τέβαλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα ενημέρωσα την Επιτροπή εκ των προτέρων ότι έχω ορισμένε αντιρρήσει για ορισμένα τμήματα τη ε, έκθεση, αλλά θα συμφωνήσω με τα άλλα τμήματα τη έκθεση. Γι' αυτό α μην συνεχίζουμε τη συζήτηση όλο το βράδυ. Ο κ. Άλβαρο ρώτησε για το αίτημα πρόσβαση από τα εθνικά DPAs. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά όταν ήμασταν στι ΗΠΑ το Φεβρουάριο, μα ενημέρωσαν ότι τίποτα δεν είχε ακόμα σταλεί ε, ως εκείνη τη στιγμή στην Αμερική. Μέσα Φεβρουαρίου λοιπόν ε, δεν είχαν ακόμη. Ίσως ε, τώρα έχουν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είχαν λάβει. Ως προς το ρόλο του JSB, Νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σύγχυση μεταξύ των δύο εκθέσεων. Υπάρχει επίσημη κοινή έκθεση που γίνεται εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το άρθρο 13 ε, τη έκθεση του FTP που δημοσιοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου. Πέραν αυτού υπάρχει η έκθεση επιθεώρησης του GSP και ναι, αυτό μπορεί να δημιουργεί σύγχυση, αλλά το GSP είναι μια ανεξάρτητη αρχή που συγκροτήθηκε από τον Ευρωπαίο νομοθέτη για να αποπτεύει όλο το έργο της Europol που έχει σχέση με τα δεδομένα και την προστασία των δεδομένων. Συνεπώς, από την αρχή του, της συμφωνίας GSDP, ο ρόλος της Europol ήταν σαφής και ε, το εποπτικό όργανο αποφάσισε ήδη το Σεπτέμβριο ότι θα γίνει μια πρώτη επιθεώρηση το ταχύτερο δυνατόν και τελικά έγινε στις 11 Νοεμβρίου και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα είναι η τελευταία επιθεώρηση. Θα ε, συνεχιστούν οι επιθεωρήσεις και από ό,τι άκουσα από την κυρία Ρέγμορτ σήμερα και από ό,τι βλέπω στο έγγραφο είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις και θα συνεχιστεί η συζήτηση των βελτιώσεων με την Europol στις μικτές συνεδριάσεις. Ευχαριστώ. Thank thank We We our guest speakers here. them. Ευχαριστούμε τους προκλημένους. If you let me, Mrs. Ludford, I just want to, for the time being, just thank θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, γιατί κάθισαν ε, περισσότερο. We should fast forward και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτό το θέμα είναι αμφισβητούμενο, είναι ένα θέμα που δημιούργησε αμφιγνωμίες από την αρχή της θητείας μας. Έτσι είχε και έτσι έχει. Άρα αν θέλετε κάτι, ένα τελευταίο σχόλιο. Έχουμε όμως άλλο ένα θέμα, κυρία Λάντφορ. Χρήσιμη αυτή η συνεδρίαση, αλλά δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το ότι υπάρχει αυτή η διαφωνία μεταξύ της κοινή εποπτικής αρχής Κομισιόν και Europol. Ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Βάιτσπορτ, είπε ότι διαφωνεί Σε ποιο τμήμα της αναθεώρησης αναφέρεται δεν μπορούμε να δίνουμε άφεση αμαρτιών συνέχεια. Συμφωνώ με τον κύριο Μπουζούτιλ κατά πολέμηση της τρομοκρατίας ζω στο Λονδίνο. Αρκεί να σας πω αυτό. Αλλά αυτή δεν είναι καλή βάση ε, εργασίας. Θα πρέπει να βρούμε μία άκρη. Can you,